Good morning, dear colleagues. Uh, uh, Γεια σας, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη μέρα της συνεδριάς της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Ξεκινώ μια ανακοίνωση κατόπιν ετοίματος της κυρίας Γκάμπρελ της ηγήτριας στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης σημερινής συνεδρίασης η απελευθέρωση των θηρήσεων με τη Γεωργία αναβάλλεται για τη συνεδρίαση της Δευτέρας 25ης Απριλίου, δηλαδή την επόμενη Δευτέρα. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ευρωπαϊκά ταξιδιωτικά γραφεία για την επιστροφή υπηκών τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα. Θα δώσω το λόγο να παρουσιαστεί το σχέδιο εκθέσεως στον εισηγητή μας, ο οποίος θα μας κάνει μια παρουσίαση του θέματος. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Μία από τις μεγάλες αποτυχίες της ευρωπαϊκής κοινής πολιτικής ασύλου και της κοινή προσέγγισης για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν καταφέρει να επαναπατρίσουν τους μετανάστες εκείνους των οποίων η αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί και που δεν χρειάζονται διεθνή προστασία και που χρησιμοποιούν τη διαδικασία χορηγήσεως ασύλου σαν δίωδο οικονομικής μεταναστεύσεως. Λιγότερο από 40% των αποφάσεων για επιστροφή και εφαρμόζονται. Αυτή η αποτυχία, η οποία έχει πολλές συνέπειες. Πρώτα απ' όλα ενθαρρύνει την κατάχρηση του συστήματος ε, ασύλου. Γνωρίζουμε ότι ένας μεγάλος αριθμός αυξανόμενος εκείνων που διασχίζουν τη Μεσόγειο προέρχονται από χώρες ε, οι πολίτες των οποίων είναι πολύ απίθανο να θεωρηθούν ως πρόσφυγες. Υπονομεύεται μετά και η εξοπιστία του συστήματος ασύλου στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο είναι ότι απορροφά πόρους που θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται προς όφελος εκείνων που πραγματικά χρήζουν προστασίας. Οι λόγοι πίσω από το χαμηλό ποσοστό επιστροφών είναι περίπλοκοι και σαφώς δεν υπάρχει μια μοναδική μαγική λύση στο πρόβλημα. Κάποια κράτη-μέλη είναι πιο επιτυχή από άλλα όσον αφορά τον επαναπατρισμό των ανθρώπων σε κάποιες χώρες καταγωγής. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να ερευνήσουμε εκ του σύνεγγυς τις διάφορες εμπειρίες και πρακτικές των κρατών μελών. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση, υπάρχουν όμως διάφορα μικροπράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ένας λόγος που έχει εντοπιστεί για το δισταγμό κάποιων χωρών καταγωγής να δεχτούν τους πολίτες τους όταν επαναπατρίζονται είναι η έλλειψη εναρμονισμένου εγγράφου ενιαίας χρήσεως με χαρακτηριστικά ασφαλείας που θα αναγνωρίζεται και από τις χώρες προέλευσης. Η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπής προσπαθεί αυτό το θέμα να το διευθετήσει υποστηρίζω ε, κατά πολύ αυτή την πρόταση με έναν αρμονισμένο ταξιδιωτικό έγγραφο ελπίζουμε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και τις δαπάνες όχι μόνο για μας αλλά και για τις ε, εμπλεκόμενες τρίτες χώρες. Οι προτάσεις μας συμπεριλαμβάνουν την ανάγκη να εξασφαλίζουμε πιο υψηλά επίπεδα τεχνικά και ασφαλείας όσον αφορά την ε, προφύλαξη έναντι πλαστογράφησης των γράφων αυτών Γι' αυτό πέραν από άλλες από άλλα προτινόμενα χαρακτηριστικά ασφαλείας των εγγράφων προτείνω να θέσουμε τεχνική προδιαγραφή για την φωτογραφία η οποία θα εμφανίζεται επί του εγγράφου αυτού. Αυτό το αναθεωρημένο ταξιτικό έγγραφο δεν αναφορά μόνο τα αυξημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, είναι και θέμα δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τρίτων χωρών. Γι' αυτό πρότεινα το εξής όπου είναι απαραίτητο και είναι διαθέσιμο αυτό να διατίθενται περαιτέρω ε, πληροφορίες για ένα άτομο ε, που αφορούν την διακίνηση ανθρώπων κλπ. Γι' αυτό προτείνω το έγγραφο να εκδίδεται σε επίσημη γλώσσα του κάτους μέρους που εκδίδει το έγγραφο, καθώς και στα αγγλικά ή γαλλικά και μια επίσημη γλώσσα της εμπλεκόμενης τρίτης χώρας. Κυρία Πρόεδρε, δεν θα πρέπει να αφήσουμε να περάσουν τα χρόνια όπως πριν, πριν καλύψουμε τα κενά στη συνεργασία μας με τρίτες χώρες ή ε, όσον αφορά τα έγγραφα που εκδίδουμε. Ε, γι' αυτό προτείνω τακτικά και διεξοδικά να αναλύουμε και να αναθεωρούμε ε, το πώς χρησιμοποιείται και πώς χρησιμοποιείται αυτό το έγγραφο, το και ποιο είναι το ποσοστό να στον των λογοταξιδιωτικού εγγράφου από τρίτες χώρε. Τέτοια στοιχεία θα μα δώσουν μια σαφή εικόνα. Θα ξέρουμε πού βρίσκονται διάφορε αδυναμίε προς διόρθωση. Δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό τα ποσοστά επιστροφή εξαρτώνται πράγματι από το ταξιδιωτικό έγγραφο. Όλο και περισσότερο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και οι δυνάμεις της τάξης αναφέρονται στην ανάγκη για διαλειτουργικότητα όσον αφορά τα συστήματα πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και την ανάγκη η πληροφορία να μην απομονώνεται σε διάφορα στεγανά, αλλά να υπάρχει επικοινωνία για να έχουμε πλήρη εικόνα όσον αφορά την κατάσταση που αντιμετωπίζεται και τι είδου δράσεις απαιτούνται. Για να αυξήσουμε λοιπόν την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων περί ασύλου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και για να αποφύγουμε δευτερογενείς μετακινήσεις τον άσυλο που, έχουν, που έχει απορριφθεί η αίτησή τους, θα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών. Είναι ουσιαστικό αυτό σχετικά με την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων και ποια άτομα θεωρούνται υπήκοοι των χωρών που διαμένουν παράνομα. Γι' αυτό προτείνω τα αντίγραφα των εγγράφων που εκδίδονται από τα κράτη-μέλη να μπαίνουν στο σύστημα Eurodac και στο σύστημα πληροφοριών Schengen. Τέλος, ούτως ώστε αυτό το έγγραφο να αναγνωρίζεται ευρέως και να είναι αποτελεσματικό, θα ήταν αναγκαίο αυτό να αποτελεί ένα κομμάτι πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πιο αποτελεσματικές συμφωνίες επανεισδοχής με τρίτες χώρες. Η αναγνώριση του εγγράφου θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενο για η αδίποτε μελλοντική συμφωνία συνεργασία και επανεισδοχή. Κυρία Πρόεδρε, η μετανάστευση είναι ευαίσθητο ε, θέμα με, πολύ, με πολλές πολιτικές αποχρώσεις. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να τονίσουμε ότι αυτή η πρόταση δεν αφορά την αλλαγή των κανόνων ή την θέσπιση νέων. Αφορά την καλύτερη εφαρμογή και επιβολή των κανόνων εκείνων που ήδη ισχύουν. Αυτό πιστεύω θα ήταν ε, επωφελές ε, για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λάχου. Και τώρα θα ξεκινήσει ο διάλογος, θα μιλήσουν σκιώδεις ηγητές καταρχάς. Η κυρία Μουσολίνη, α δεν τη βλέπω, την είδα πριν αλλά δεν είναι εδώ. Η κυρία Ντάτη λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για τις προτάσεις του για αυτό το νομοθετικό θέμα. Οι σοσιαλδημοκράτες πιστεύουμε ότι μια προσφυγική πολιτική, μια μεταναστευτική πολιτική η οποία να είναι λειτουργική απαιτείται για να το πετύχουμε να ληφθούν μέτρα που να καλύπτουν όλα τα φαινόμενα τα οποία αυτή τη στιγμή εκδηλώνονται. Από την άφηξη από την αναχώρηση μάλλον από τη χώρα καταγωγής, όπως επίσης και την επιστροφή τους. Θα πρέπει να βλέπουμε το σύνολο της εικόνας, χορηγώντας ή αρνώντας ε, το άσυλο μόνο, αρνούμενη συγγνώμη το άσυλο μόνο, δεν είναι κάτι το οποίο ε, θα δώσει λύση. Το 60% υποτίθεται των μεταναστευομένων ε, θα πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες τους, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούν να ζουν στη χώρα υποδοχής κάτω από απαράδεκτες συνθήκες, σε πλήρη φτώχεια και χωρίς καμία εγγύηση. Έχουν ε, εμπλακεί σε μια κατάσταση νομικής ανυπαρξίας γιατί οι χώρες τους ε, δεν δέχονται να τους υποδεχθούν λόγω έλλειψης εγγράφων ή γιατί δεν αναγνωρίζουν τα έγγραφα τα οποία έχουν. Ε, είναι σωστό βέβαια αυτό, όχι, αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο είναι κατά και τη άρθρο 13 της Συμφωνίας του Κοτονού. Ακριβώς η πρόταση αυτή προσπαθεί να δώσει μια απάντηση στο συγκεκριμένο θέμα, διασφαλίζοντας ε, με ένα ξεκάθαρο κείμενο το οποίο θα διευκολύνει την αποδοχή από τις χώρες και ταυτόχρονα θα διασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών. Είναι ένα τεχνικό θέμα και δεν θα δεχθούμε επιπλέον προσθήκες που θα θέσουν σε κίνδυνο τους ανθρώπους αυτούς όταν επιστρέφουν στην χώρα τους, γιατί οι επιστροφές είναι τμήμα της μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά θα πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μεταναστών. Ε, ελπίζουμε λοιπόν ότι θα συνεισφέρουμε περαιτέρω και θα καταλήξουμε σε ένα νομοθετικό φάκελο ο οποίος θα μπορέσει να βρει λύσεις. Ευχαριστώ κυρία Ντάλη, κυρία Μουσολίνη. Πρόεδρε, εμείς σαν πολιτική ομάδα συμφωνούμε απολύτως πάνω στο έγγραφο αυτό. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό είναι ένα έγγραφο το οποίο ανανεώνει το παλαιό του 1994 και από το 1994 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά, έχουμε περάσει πολλές κρίσεις. Τώρα δεν μιλάμε για μία απλή κρίση, αλλά μιλάμε για ένα χρόνιο πρόβλημα. Η θέση μας για το σύνολο της έκθεσης είναι θα έλεγα ευνοϊκή. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να εντάξουμε ε, στην πρόταση αυτή είναι κάποιες διευκρινήσεις γύρω από τις ε, συμφωνίες επανεισδοχής. Να δοθεί δηλαδή μεγαλύτερος ρόλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συμπροταγωνιστικό ρόλο με τα κράτη-μέλη τα οποία δρούν επιτόπου στα πλαίσια της ανάλυσης ε, και των αναγκών που υπάρχουν για τα συγκεκριμένα έγγραφα. Γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι δεν ασχολείται η πρόταση με τις συνθήκες ε, ε, επαναπατρισμού, αλλά είναι ένα τεχνικό ε, έγγραφο το οποίο θα προσπαθήσει να προχωρήσει στην περαιτέρω τυποποίηση αυτού του είδους των εγγράφων. Αυτό το οποίο είναι το βασικό λοιπόν είναι να, υπάρξει, να υπάρξουν διευκρινήσεις, να είναι ξεκάθαρο το κείμενο και σε επίπεδο διατύπωσης και σε επίπεδο τεκμηρίωσης. Είναι ένα τεχνικό όπως είπα έγγραφο, δεν πρέπει να δημιουργούνται παρανοήσεις, αντιφάσεις, γιατί πλέον σε επίπεδο διμερών σχέσεων το παλαιό κείμενο δεν γίνεται δεκτό. Πρέπει λοιπόν να είναι σαφές το κείμενο αυτό και δεν πρέπει να αγνοεί τις αλλαγές που έχουν επέλθει στον τομέα αυτό. Πρέπει να υπάρξει επίσης και αναφορά στους ε, μη ε, συνοδευομένους ανηλίκους σε συγκεκριμένο παράρτημα. Και θα πρέπει επίσης να δούμε και τι επιπλέον οικονομικά βάρη προκαλεί η ιστορία αυτή ε, στα κράτη τα οποία θα πρέπει να εφαρμόσουν τον κανονισμό. Ευχαριστώ κυρία Μουσολίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Σιγητά. Οι παράνομοι μετανάστες που αρνούνται να επιστρέψουν είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και δεν είναι μυστικό ότι το πρόβλημα αυτό θα ε, γίνει μεγαλύτερο στο μέλλον πολλές φορές ε, συνδέεται ε, αυτό με εγκληματικότητα και πρέπει να τηρηθεί ο νόμος διότι διαφορετικά υπονομεύεται το κράτος δικαίου. Είναι ένα αναγκαίο κακό θεωρώ διότι οι επιπτώσεις ε, της μη επιστροφής είναι τεράστιες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν χαιρετίζω την πρόταση του εισηγητή και συμφωνώ με την τροπολογία 5α, τη, η αναγνώριση αυτών των νέων ε, ταξιδιωτικών εγγράφων θα πρέπει να είναι προϋπόθεση για ε, ένα τρίτο κράτος ε, μέλος. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Βίμπερ και κυρία Σαρτζεντίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και συγγνώμη για την αργοπορία. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι μια και το θέμα είναι τεχνικό, καλύτερα θα ήταν να παραμείνει τεχνικό, διότι διαφορετικά δεν θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε εάν μετατρέψουμε το τεχνικό σε πολιτικό ζήτημα. Τουλάχιστον ε, αυτό θεωρούν οι πράσινοι. Δεν νομίζω ότι προσπαθώντας να επιστρέψει κάποιος στη χώρα του αφού έχει αρνηθεί το αίτημα ασύλου, έχει να κάνει με προβλήματα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τρίτη χώρα πρέπει να επιτρέψει την επιστροφή του ατόμου αυτού. Και έχω δει περιπτώσεις ανθρώπων που θέλουν να γυρίσουν πίσω, αλλά η χώρα τους δεν τους αναγνωρίζει και δεν μπορούν να λάβουν τα, τα κατάλληλα έγγραφα. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα, ό,τι και αν κάνουμε από την πλευρά μας. Το δικό μου λοιπόν ερωτηματικό είναι γιατί επιθυμούμε κάτι ε, τέτοιο, να λες επασέρ, διότι μία χώρα που θέλει να δεχτεί πίσω έναν υπηκό της θα του έδινε τα κατάλληλα ταξιδετικά έγγραφα. Εάν θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να διευκολύνουμε τη διαδικασία των επιστροφών, σε περίπτωση βέβαια που ε, όσοι επιστρέφονται γίνονται δεκτοί από, το τρίτο, από την τρίτη χώρα, ε, καλώς. Όμως, εάν σκοπεύουμε με αυτό να μετακινούμε τους ανθρώπους αυτούς από χώρα σε χώρα, νομίζω πως δεν έχει κανένα νόημα, διότι δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Αν δεν θέλεις κάποιον στη χώρα σου δεν υπάρχει περίπτωση να ε, τον πάρεις πίσω. Γι' αυτό καταλαβαίνω και τις ε, επιπλέον αιτιολογικές σκέψεις του εισηγητή που ε, έχουν να κάνουν με την πολιτική του τοποθέτηση. Δεν τις συμμερίζομαι βέβαια, όμως πιστεύω πως αυτές οι επεξηγήσεις βοηθούν στην κατανόηση αυτού του τεχνικού θέματος. Για παράδειγμα, αυτό το έγγραφο θα έχει φωτογραφία και μας ε, λέει ο εισηγητής πως η φωτογραφία θα είναι τύπου διαβατηρίου. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι λογικό και ότι εντάξει καλύτερα να έχεις μια φωτογραφία τύπου διαβατηρίου παρά μια φωτογραφία από τις διακοπές κάποιου στην παραλία. Πώς όμως θα βγάλεις αυτή τη φωτογραφία όταν κάποιος δεν είναι στο σύστημα, δεν θέλει να φωτογραφηθεί διότι δεν θέλει να τον απελάσουν, πώς θα καταφέρουμε να βγάλουμε αυτή τη φωτογραφία. Αυτές είναι λεπτομέρειες τις οποίες ε, πιστεύω χρειάζεται να διευκρινίσουμε. Θα μείνω εδώ, κύριε Πρόεδρε, ακριβώς γιατί άργησα, όμως θα ήθελα να κάνω άλλη μια φορά έκκληση να μην μετατρέψουμε το θέμα σε πολιτικό, να μην αρχίσουμε να συζητάμε την πολιτική επιστροφών, διότι έτσι δεν θα καταφέρουμε ποτέ να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βεζιά, θέλετε να πάτε το λόγο, Σκιώθης. Συγγνώμη, έφτασα καθυστερημένα. Θέλω να πω ότι δεν εκπλήσωμαι που βλέπω την εκδοχή αυτή ε, του κειμένου Συμφωνώ την κυρία Σαρτζεντίνη. Το θέμα αυτό πρέπει να παραμείνει τεχνική φύσεω, αν θέλουμε να προχωρήσουμε και όχι πολιτικό εργαλείο. Λυπάμαι για την καμπή που παίρνει το όλο ζήτημα. Ευχαριστώ κυρία Βερζιά. Άλλο μέλο που θα ήθελε να παρέμβει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάτι να προσθέσει. Ορίστε. Καλημέρα σε όλους σας. Εμμανουέλ Καμπό είναι το όνομά μου από την DG Home να πω κάποια πράγματα για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο λόγος υποβολής προτάσεως είναι εξή. Για την ώρα δεν έχουμε ένα αρμονισμένο έγγραφο επιστροφής με ισχυρά χαρακτηριστικά ασφαλείας και ξέρουμε ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα. Κάτι που επηρεάζει την πολιτική επανεισδοχή που θέλουμε να γίνει πιο αποτελεσματική και είναι προτεραιότητα Ευρωπαϊκή Ενώση και κρατών μελών. Τι προσπαθούμε μέσω τη προτάσεω θέλουμε εντός της αλυσίδας επανεισδοχής να εξασφαλίζουμε ότι τα αξιωτικά έγγραφα αποτελούν ισχυρό στοιχείο. Δεν θέλουμε να έχουμε ένα αδύναμο στοιχείο εδώ όπως κατά το παρελθόν, διότι κάποιες χώρες δεν δεχόταν τα ταξιδιωτικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ενώσης διότι δεν είχαν επαρκή χαρακτηριστικά ασφαλείας. Θέλουμε λοιπόν να ισχυροποιήσουμε ένα στοιχείο της αλυσίδας. Με την πρόταση αυτή δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα που αφορούν την επανεισδοχή και ξέρουμε ότι έχουμε αρκετά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Είναι τεχνική φύσεως πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ένα αξιόπιστο έγγραφο ε, ταξιδιωτικό επιστροφής και δεν μπορούμε να το μετατρέψουμε σε κάτι άλλο. Κάποια σχόλια ή Κάποιες τροπολογίες αφορούν τα τεχνικά πρότυπα για τη φωτογραφία, μετάφραση, πληροφορίες, περισσότερες πληροφορίες. Πρέπει να μελετήσουμε τις προτάσεις προσεκτικά, ούτω ώστε να μην γίνει πιο επαχθής η διαδικασία, να μην αυξάνει τη γραφειοκρατία και να καταλήγουμε σε προστιθέμενη αξία μέσω αυτών. Διότι το ταξιδιωτικό έγγραφο πρέπει να είναι εύχριστο για τα κράτη-μέλη και δεν θα πρέπει να είναι ακριβό αν θέλουμε να χρησιμοποιείται. Τώρα για τις τροπολογίες που αφορούν το άρθρο 5α για να εξατάται η συμφωνία επανεισδοχής από τη χρήση του αξιωτικού έγγραφου, αν το κάνουμε αυτό θα είναι αντιπαραγωγικό να υπάρχει αυτή η συνάρτηση. Είναι πολύ δύσκολες οι διαπραγματεύσεις με τις χώρες επανεισδοχής. Κάποιες από αυτές δεν θέλουν να δεχθούν μια συμφωνία επανεισδοχής, άρα χρειαζόμαστε μια ευκαμψία και αυτό απαιτεί συνεχείς πολιτικές προσπάθειες. Δεν θέλουμε να υπάρχει αυτός ο σχετισμός, θα ήταν αντιπαραγωγικό για τις θεωρήσεις. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούσαμε κάποιο στοιχείο μόχλευσης και με κάποια κράτη, με κάποιες χώρες, τρίτες χώρες που δεν συνεργάζονται για επανεισδοχή, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το μοχλό πίεση τη θεωρήσεω και το συζητούμε αυτό με τα κράτη-μέλη. Για την ώρα αναδιατυπώνεται όλος κώδικα για τις θεωρήσει είναι στον τριμερή διάλογο η διαδικασία. Θα πρέπει αυτό να το συζητήσουμε στα πλαίσια του κώδικα για τις θεωρήσεις. Εδώ η συγκεκριμένη πρόταση δεν είναι ο κατάλληλο χώρος για αυτού του είδου συζητήσει, για το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν και το Eurodac. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν και ενδεχομένω και το Eurodac, ούτω ώστε να έχουμε πληροφορίε ε, από πλευρά κατών μελών για τι αποφάσει επιστροφή. Και γίνεται μελέτη σκοπιμότητα να δούμε κατά πόσο στην απόφαση περί επιστροφή μπορούμε να συμπεριλαμβάνουμε πληροφορίε και αυτέ οι πληροφορίε να είναι στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη σκοπιμότητα, υπάρχουν κάποιε δυσκολίε διότι στο σύστημα πληροφοριών Schengen και στο Eurodac μπορούμε να εισαγάγουμε κάποια στοιχεία αλλά όχι ένα έγγραφο. Πρέπει να δούμε τι είναι εφικτό και μετά από τη μελέτη σκοπιμότητας ίσως να υπάρξει πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά εδώ δεν είναι το κατάλληλο πλαίσιο να συζητήσουμε αυτό το θέμα όταν συζητάμε το έγγραφο. Τι θέλω να πω. Προσπαθούμε να εξετάσουμε ένα τεχνικό ζήτημα και πρέπει να περιοριστούμε σε αυτό το πλαίσιο. Διότι αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι να έχουμε ένα έγγραφο που θα εγκριθεί το ταχύτερο δυνατόν. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καμπό. Το λόγο ξανά τον έχει ο εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω επί της ουσίας. Να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 24 Απριλίου και θα προσπαθήσουμε να διοργανώσουμε την επόμενη συνεδρίαση των σκιωδών. Μου λένε 28 Απριλίου, λέει η Πρόεδρος, 5 το απόγευμα η προθεσμία της τροπολογίας. Έκανα λάθος, λέει ο συγγητής, ζητώ συγγνώμη. Καλώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε συγγητά. Πάμε στο επόμενο σημείο. Ενίσχυση των ελέγχων και συγκρίσεων βάσεων δεδομένων ε, σχετικά με τα εξωτερικά σύνορα. Η κυρία Μακοβέ είναι εδώ που είναι η συγγήτριά μας. Είναι σημαντικό το η πρόταση. Θα σας δώσω αμέσως το λόγο, κυρία η συγγήτρια. Κυρία Μακοβέ έχει το λόγο. doamna președintă. Um, securitatea și Ευχαριστώ πρόεδρε. Η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών είναι για μας η απόλυτη προτεραιότητα. Οι περισσότεροι από τους Ισλαμιστές που τομοκρατούν τους Ευρωπαίους είναι πολίτες της Ευρώπης. Και το φαινόμενο της τζιχάντ έχει πάρει ε, θα έλεγα τεράστιες διαστάσεις και πρέπει να ενισχύσουμε έτσι τα εξωτερικά σύνορα και να έχουμε τα μέσα για να το πετύχουμε. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τραποποίηση του κώδικα Σέγγεν ε, επιφέρει ε, αλλαγές σε επίπεδο συστηματικό στα πλαίσια των κανόνων παρακολούθησης και των Ευρωπαίων πολιτών και των πολιτών οι οποίοι δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο βαθμό που η συστηματική αυτή έλεγχη θα δημιουργήσουν προβλήματα στο πέρασμα των συνόρων, σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να κάνουν επιλεκτικούς ελέγχους, τυχαίους ελέγχους, επί τη βάση της αξιολόγησης του κινδύνου, την οποία θα κάνει η συγκεκριμένη υπηρεσία. Μια τέτοια αξιολόγηση θα πρέπει να αποδεικνύει ότι οι έλεγχοι αυτοί θα έχουν συγκεκριμένους στόχους Ποια είναι τώρα τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της έκθεσης αυτής, θα σας τα παρουσιάσω συνοπτικά βέβαια. Υπάρχουν κάποιες νέες προτάσεις σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν εξαιρέσεις για, αυτούς τις, για αυτές τις μορφές ελέγχου. Όπως είπαμε βασίζονται σε αξιολογήσεις κινδύνου για μια περιορισμένη χρονική περίοδο. και για όλα τα είδη των συνόρων, θαλάσσια και τα λοιπά, ε, υπηρετικά επίγεια και τα Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν προσαρμογές έτσι ώστε να επανέλθει στο κανονικό η κυκλοφορία των πολιτών στα σύνορα. Οι εξαιρέσει μπορεί να είναι περιορισμένες στο χρόνο, σε μια πρώτη φάση έξι μήνες μετά από τη θέση σε ισχύ του νέου κανονισμού. Από αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι αυτή η προθεσμία των έξι μηνών είναι, μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλη και γι' αυτό θα προτείνω μια μικρότερη περίοδο σχετικά τώρα με την αξιολόγηση των κινδύνων. Οι εξηγήσει αυτές θα πρέπει να δίδονται όχι μόνο στη Frontex αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις όμορες χώρες. Σε μια άλλη τροπολογία μου προτείνω ότι 12 μήνες μετά τη θέση σε ισχύ του κανονισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μεταφέρει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μια αξιολόγηση των συνεπειών αυτής της εξαίρεσης από τους κανονικούς κανόνες. Θα πρέπει λοιπόν το κόστος <clears throat> σε επίπεδο πρακτικό των ελέγχων αυτών να είναι το ελάχιστο δυνατό. Θα πρέπει επίσης να αποφευθεί η επικάλυψη των ελέγχων, ο διπλός έλεγχος για αυτούς οι οποίοι περνούν τα σύνορα. Εδώ τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν ελέγχους στο έξοδο, στην έξοδο της χώρας. <clears throat> Στόχος αυτής της εξαίρεσης είναι να αποφευθούν έλεγχοι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα με βάση την ίδια βάση δεδομένων. Η χώρα μου θα προτιμούσε οι έλεγχοι αυτοί να γίνονται όσο πιο συχνά γίνεται και άλλωστε εφαρμόζουμε το κανόνα αυτό για τα εξωτερικά σύνορα της χώρας μας από τον Σεπτέμβριο του 2015. Στην τροπολογία 14 για την ενίσχυση της ασφάλειας, οι χώρες που έχουν επαναφέρει σε προσωρινή βάση τον εξωτερικό έλεγχο, λέμε να γίνεται αυτό με συστηματικότερο τρόπο, επί τη βάση των κανόνων που είναι σε ισχύ σήμερα. Θα πρέπει να ισχύει ο κανόνας μουτάντης μουτάντης για τον έλεγχο των ε, συνόρων. Η τροπολογία 22 για τη χρήση όλων των μέσων τα οποία είναι διαθέσιμα. Προτείνω ότι εκεί που κάτι τέτοιο είναι εφικτό, οι πολίτες οι οποίοι δεν έχουν την υπηκότητα του συγκεκριμένου κράτους κάθε φορά, να εντάσσονται σε μια βάση δεδομένων ευρύτερη που θα περιλαμβάνει και τους πολίτες εκτός Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οι υπηρεσίες να είναι σε θέση να ελέγχουν και επιπλέον βάσεις δεδομένων, όχι μόνο της Europol και τις εθνικές κάθε φορά. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορεί να γίνουν με βάση διμερείς συμφωνίες που έχουν υπογραφεί ανάμεσα σε χώρες και σε τρίτες χώρες της Ένωσης και σε τρίτες χώρες, όπως επίσης και σε συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεργαστεί καλύτερα σε διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση της δημοκρατίας. Συμπερασματικά, οι πρόσφατες τρομοκρατικές ενέργειες επιβεβαιώνουν ότι η συμπληρωματική έλεγχη είναι κάτι το οποίο έχουμε ανάγκη, πρέπει να δώσουμε εγγυήσεις στον Ευρωπαίο πολίτη. Υπάρχει ένα άγχος στον Ευρωπαίο πολίτη ε, λόγω των τελευταίων επιθέσεων, αμφισβητείται το δικαίωμά του στη ζωή και εγώ είχα επαφές με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών από διάφορες χώρες και όλοι είναι πεπισμένοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει ό,τι μπορεί και τα μέτρα τα οποία λαμβάνει, τα λαμβάνει ε, σε περιορισμένη βάση και εκ των υστέρων. Και από την άλλη οι τρομοκράτες είναι πάντα καλύτερα προετοιμασμένοι, προβαίνουν στις τρομοκρατικές τους ενέργειες και εμείς δεν κάνουμε παρά τίποτα από το να διορθώνουμε τις συνέπειες. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε με υψηλότερη ταχύτητα. Πρέπει να καταγγείλουμε την γραφειοκρατία η οποία μας χαρακτηρίζει. Δεν μιλάμε μόνο για τον κώδικα Σέγγεν, αλλά μιλάμε επίσης γενικότερα για το θέμα της ασφάλειας των σύνορων. Μιλάω για τα εξωτερικά κυρίως σύνορα Έτσι θα αποφύγουμε την απώλεια ανθρώπινης ζωής στο μέλλον. Περιμένω τις προτάσεις σας. Η προθεσμία ε, για τις ε, τροπολογίες είναι 23η Απριλίου. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μακοβέη. Θα δώσω τώρα το λόγο στους κύριους δισηγητές. Κυρία Κοντρίτσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μακοβέ για την ε, λεπτομερή της παρουσίαση. Στο ΡΑΚ ε. συμφωνούμε σε γενικές γραμμές με το περιεχόμενο της έκθεσης, που σημαίνει ότι οι μελλοντικέ αλλαγές, ιδιαίτερα ε, σε σχέση με την ασφάλεια στον χώρο του Σέγγεν, μας ικανοποιούν. Θεωρούμε πως ο κύριος στόχος θα πρέπει να είναι η ασφάλεια των πολιτών της Ένωσης. Επομένως, τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης πρέπει να είναι ασφαλή με τρόπο πιο αποτελεσματικό και αυτό συμπεριλαμβάνει και την ανταλλαγή δεδομένων με κατάλληλο τρόπο, φροντίζοντας πάντα την προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων. Στηρίζω επίση τη μεταβατική περίοδο των έξι μηνών για τα εναέρια σύνορα. Πιστεύω πως αρχικά τουλάχιστον δεν ε, θα έχει δυσανάλογες επιπτώσεις στο κόστος των αερομεταφορών. Πρέπει να δεχτούμε αυτήν την χρονική περίοδο των έξι μηνών ως μεταβατική. Θα υποβάλω ορισμένες τροπολογίες οι οποίες θα επιτρέψουν την πρόσβαση σε όλες τις βάσεις δεδομένων έτσι ώστε να μπορούμε να καθορίσουμε ε, το αν κάποιος απειλεί την δημόσια ασφάλεια. Επίσης, χρειάζεται να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν και να εμπλουτίζουν τις βάσεις δεδομένων. Θα ήθελα επίσης να τονίσω πόσο σημαντικό ειδικα ειναι είναι κάποια κράτη-μέλη που έχουν εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν ανήκουν ακόμα στο χώρο του Σέγγεν. Είναι πολύ σημαντικό να αλλάξει αυτό έτσι ώστε να ε, γίνουν πιο ασφαλή τα εξωτερικά σύνορα. Θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες γι' αυτό και αναμένω την Επιτροπή να παρέχει στήριξη στα κράτη-μέλη και να δημοσιεύσει μία σύσταση για τα χρονικά δια, τα μεταβατικά διαστήματα. Επίσης, συμφωνώ με την ε, διατύπωση της κυρίας Μακοβέη σχετικά με τις ε, περιοδικές αξιολογήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κοντρίτσκα. Η κυρία Φαγιών έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τη Μόνικα για την παρουσίαση της έκθεσης δίχως αμφιβολία θέλουμε την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Όμως έχω κάποιες ανησυχίες, τις οποίες θα αναφέρω εν μέρη τώρα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι προσανατολισμένη στην ασφάλεια, πιστεύω, και παραμερίζει την αρχή της αναλογικότητας. Και θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν έγινε εκτίμηση αντικτύπου, κάτι το οποίο είναι ε, συνήθως με τέτοιες περιπτώσεις. Η συστηματική έλεγχη όλων των επιβατών που εισέρχονται ή εξέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα σημαίνει και αυξημένη ασφάλεια. Οι συνοριοφύλακες αυτή τη στιγμή είναι ήδη υπερφορτωμένοι με τις ε, υποχρεώσεις του Σέγγεν και ε, των θεωρήσεων. Και όταν ήμουν εισηγήτρια για τα έξυπνα σύνορα, για τη δέσμη μέτρων αυτή, το διαπίστωσα. Πάρα πολύ συνοριοφύλακε μου είπαν ότι στις ώρες αιχμή δεν διεξάγουν συστηματικούς ελέγχους ε, θεωρήσεων μέσω του, ε, του ηλεκτρονικού συστήματος, ακριβώς επειδή οι αεροπορικέ εταιρείε και οι επιβάτες τους ασκούν μεγάλη χρονική πίεση. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με το 1 τρίτο των διελεύσεων από τα εξωτερικά σύνορα που ε, γίνονται από επικόους τρίτων χωρών. Αν δούμε τι γίνεται με τους ε, πολίτες της Ένωσης, θα παρατηρήσουμε ότι ε, αποτελούν τα δύο τρίτα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα στα σύνορα. Και θεωρώ πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αξιολόγησε παρκώς τις επιπτώσεις της εφαρμογής αυτής της πρότασης. Θεωρώ ότι η συστηματική έλεγχη σε όλους ε, με αντιπαραβολή των βάσεων ε, δεδομένων θα έχουν αρνητικέ επιπτώσει ε, στην κίνηση των επιβατών τουλάχιστον σε ορισμένα σύνορα. Για παράδειγμα τα σύνορα Σλοβενίας-Κροατίας θα έχουν δυσκολία στην εφαρμογή αυτής της πρότασης. Αυτή τη στιγμή έχουμε 250.000 διελεύσεις κάθε χρόνο, ιδιαίτερα την τουριστική περίοδο. Να μην αναφέρω την περίπτωση του Γιβραλτάρ, όπου κάθε μέρα περνάνε τα σύνορα 10.000 άνθρωποι. Αυτοί πρέπει να ελέγχονται συστηματικά. Τι σημαίνει αυτό. Εξετάζοντας την πρόταση, θεωρώ ότι οι συστηματικοί έλεγχοι θα πρέπει να διεξάγονται μόνο όταν χρειάζεται και αυτό θα πρέπει να βασίζεται σε εκτίμηση κινδύνου, δηλαδή το αντίστροφο από αυτό που προτείνει η Επιτροπή. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε ε, φυσικά σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα μπορούσαν να εξαιρούνται από αυτό οι Ευρωπαίοι πολίτες. Θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες και ελπίζω να βελτιωθεί η πρόταση. Αυτό που σίγουρα δεν χρειαζόμαστε είναι άλλον έναν κακό νόμο, ο οποίος δεν είναι ε, εφικτό να εφαρμοστεί. Σε ευχαριστώ κυρία Ταγιάννη, κυρία Ιντεφέλτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστούμε την εισηγήτρια για την παρουσίαση. Συμφωνώ με τις περισσότερες εκφραστήσεις ανησυχίες που ακούσαμε την κυρία Φαγιών. Θέλουμε μέτρα ασφαλείας όπου αυτό είναι αναγκαίο. Ναι. Θα πρέπει να είναι κάτι αναγκαίο και να κινηθούμε αναλόγως. Αλλιώς ποιος ο σκοπός. Μιλάμε για ένα μέτρο που θα έχει τεράστιο ενδεχομένω αντίκτυπο στις ε, διάφορες ροές των ταξιδιωτών. Υπάρχει έλλειψη εκθέσεως αναλύσεως επί των ταξιδιωτικών ροών. Μας είπαν ότι στο Σαλτεγκόλ για μία μέρα το δοκίμασε η Γαλλία και ήταν τόσο χάλια η κατάσταση που εγκατέλειψαν την προσπάθεια μετά από ένα 24ωρο. Αν δεν μπορεί το αεροδρόμιο de να το εφαρμόσει αυτό, πώς να περιμένουμε να το καταφέρουν αυτό κάποια άλλα αεροδρόμια. Πραγματικά πιστεύω ότι χρειάζεται η αξιολόγηση συνεπειών πριν λάβουμε δίποτε απόφαση. Αναρωτιέμαι μάλιστα γιατί υπάρχει μια τάση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστηματικά να μην συνοδεύει προτάσεις τη που υποβάλλονται εδώ από αξιολόγηση συνεπιών. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Ποιοι λόγοι κρύβονται πίσω από αυτό. Και κάτι άλλο θέλω να καταλάβω προβλέπεται παρέκκληση από συστηματικού ελέγχου από χερσαία και θαλάσσια εξωτερικά σύνορα, αλλά όχι για αεροπορικά εναέρια σύνορα του ΣΥΠΗΝ, στα αεροδρόμια. Ποια είναι η λογική μεταξύ συστηματικών ελέγχων και εξαιρέσεων, όπου η εξαίρεση είναι η δειγματοληπτική έλεγχη, σύμφωνα με τον κίνδυνο. Αν κάτι βασίζεται επί κινδύνου, τι κάνεις, κάνεις αυτό που θέλεις να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο. Ότι δεν αποτελεί κίνδυνο, γιατί να ελέγχεται συστηματικά. Γιατί να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Ο κανόνας πρέπει να έχουμε, να έχουμε ελέγχους βάση κινδύνου και η εξαίρεση να είναι η συστηματική έλεγχη. Πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας τώρα. Έχουμε τα στοιχεία PNR, το API. Μου είπαν ότι κάποια κράτη-μέλη ασκούν πιέσεις τους μεταφορείς να συλλέγουν συστηματικά στοιχεία API και για πτήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό παραβιάζει την ομοθέσια. Πρέπει να ερευνηθεί. Πρέπει να ελέγξουμε ποια μέσα έχουμε ήδη στη διάθεσή μας και να συγκρίνουμε με τη νέα πρόταση για το σύστημα εισόδου-εξόδου. Τέλος, δύο παρατηρήσεις. Αν κάνουμε ελέγχους βάση κινδύνου, ποια θα είναι η βάση για την αξιολόγηση του κινδύνου. Ε, μια γενική εικόνα για τον κάθε άνθρωπο που, για τον οποίο μπορεί να υπάρχουν υπόνοιες. Ε, ας μην χάσουμε τα πάντα, ας απομακρυνθούμε λίγο να δούμε τη γενική εικόνα. Θέλουμε ασφάλεια. Πρέπει να αξιολογήσουμε προσεκτικότατα από πού προέρχονται οι απειλές. Τίνουμε να ελέγχουμε τους έξωθεν κινδύνους. Είναι η ανθρώπινη φύση. Να έχουμε αυτό το αντανακλαστικό. Πάντα είναι κάτι ξένο, εξωτερικό κίνδυνος. Αν δούμε τις πραγματικές απειλές που υφίστανται, όπως τις επιθέσεις, τις πρόσφατες, βλέπουμε ότι προήλθαν έσωθεν και όχι έξωθεν. Χρειάζονται μέτρα ασφαλείας, ναι. Όμως, αναλογικά, να είναι απαραίτητα και πάνω από όλα τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά. Ευχαριστώ κύριε Ντεφέλντ. Η κυρία Βεργιά έχει το λόγο. Με τη σειρά μου ευχαριστώ. την συγγήτρια Σημερίζομαι εν γέννη τις αναλύσεις που ακούσαμε της κυρίας Φαγιών και της κυρίας Ιντφελτ. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε την ασφάλεια όλων εκείνων που ζουν στην επικράτεια. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι ενθερμό αντιδράσεις ε, δεν είναι και οι πιο υγιής, Το είδα μετά τις επιθέσεις στο, στη Μαδρίτη το κείμενο της τηλεπικοινωνίες που ακυρώθηκαν αυτά τα κείμενα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Λέει η συγκήτρια στην εισαγωγή ότι πρέπει να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες από τους τρομοκράτες, άρα να ενισχύσουμε τα εξωτερικά σύνορα. Ποια λογική ακολουθείτε. Δεν καταλαβαίνω το επιχείρημα. Έχουμε μία μανία με τους ελέγχους όλων των πολιτών, όλων εκείνων που καταφθάνουν στην επικράτειά μας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό χωρίς να επηρεάσουμε τις ροές, χωρίς να αυξηθεί ο χρόνος αναμονής στα σύνορα. Δεν κατανοώ. Πρέπει να το ομολογήσω αυτό. Πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς αύξηση του κόστους. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση το καταλαβαίνω, αλλά για τα κράτη-μέλη δεν νομίζω να μην υπάρξει αύξηση του κόστους. Χρειάζονται ανθρώπινοι πόροι. Αν θέλουμε να αποφύγουμε ουρές. Προτείνεται καλύτερη συνεργασία με το εξωτερικό. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να επιβάλλουμε σε ένα ευρωπαϊκό κείμενο στις τρίτες χώρες να κινηθούν όπως τα κράτη-μέλη. Ε, είναι απλώς ευχολόγιο αυτό. Και έχω ερωτηματικό επ' αυτού. Όλοι ξέρουμε ότι το πρόβλημα στην πραγματικότητα είναι η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Η κυρία Φαγιού ανέφερε παραδείγματα. Το ίδιο για την αναλογικότητα. Μελέτε συνεπιών αντιχτύπου που είναι απαραίτητες. Η Σοφίντ Βέλτ αναφέρθηκε στο Σαλ Γκολ εγώ θα πάρω ένα μικρό αεροδρόμιο σαν παράδειγμα. Το Στρασβούργο. Όταν προσπάθησαν να εφαρμόσουν εκεί στο Στρασβούργο, στο Στρασβούργο στο αεροδρόμιο συστηματικούς ελέγχου ήταν φρικτή κατάσταση. Διότι δεν είχε τα μέσα το αεροδρόμιο του Στρασβούργου να εφαρμόσει αυτού του είδους ελέγχους. Και αν το κάνει, καλή τύχη εύχομαι. Εγώ παίρνω το τρένο, δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Καλή τύχη εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους όμως που καταθάνουν αεροπορικός ή Στρασβούργο. Θα πρέπει να προβλέψουν συμπληρωματικό χρόνο αναμονής κατά την άφηξη και κατά την αναχώρηση. Προσθέτω ότι μέχρι τώρα τα κράτη-μέλη πάντα είχαν τη δυνατότητα συστηματοποίησεως των μεθοριακών ελέγχων Σέγγεν μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι Ιανουάριο και Νοέμβριο του 2015 ζήτησε συστηματικού ελέγχους η Γαλλία και αυτό δεν πραγματοποιήθηκε. Σήμερα τοποποιούμε τον κανονισμό Σέγγεν για να αντιστρέψουμε το βάρος της απόδειξης θα έλεγα εγώ. Δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό θα αλλάξει οτιδήποτε. Δεν αποτελεί επανάσταση. Τα κράτη-μέλη για μία ακόμη φορά απευθύνονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλυφθούν τα κενά τους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ένωση απαντά με συμπληρωματικά κείμενα. Νομίζω ότι δεν προχωράμε, δεν κάνουμε τίποτα. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η συνοχή όλων αυτών. Διότι θέλουμε να τροποποιήσουμε όλα τα κείμενα όσον αφορά τον τομέα αυτό. Πώς θα διαθροθεί αυτό, πώς θα συντονιστεί Τούν αυτά με τα κείμενα που εγκρίναμε το PNR, με το κείμενο που θα εξετάσουμε ε, για τα ευφυή e σύνορα, έχουμε και ένα έντυπο για το Eurodac, όλα αυτά πώς θα συντονιστούν. Δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω πια όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τι κάνουμε. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη, το επαναλαμβάνω, προσπαθούν να απαλλαχθούν, να απεμπολίσουν τις ευθύνες τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μια διακριτή προσωπικότητα ξεχωριστή από τα κράτη-μέλη. Να θέτουμε επί χάρτου ευθύνε που θα αναθέτουμε στι αρχέ Ευρωπαϊκή Ενώσεω είναι κάτι που, που δεν είδε θα διευθετήσει το πρόβλημα των συμπολιτών μα και όλων εκείνων που ζουν στην επικράτειά μα. Βέβαια είμαι λίγο προκλητική. Δυστυχώ φοβούμαι ότι δεν μπορούμε να εμποδίσουμε επόμενη απόπειρα, επόμενη επίθεση και περιμένω τι θα μα προταθεί τότε σαν νέο μέτρο ε, που θα, ε, δεν θα υπονομεύει και τις ελευθερίες μας. Ευχαριστώ κυρία Βερζιά. Η ε, κυρία Λούνατσεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μακοβέη για την παρουσίασή της. Να πω και εγώ ότι συμμερίζομαι τις ανησυχίες που έθεσαν οι τελευταίοι ομιλητές. Το θέμα της ασφάλειας είναι βασικό. Αλλά απαιτείται αναλογικότητα, αναγκαιότητα και αυτό δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι τώρα από την Επιτροπή. Και αυτή είναι και γνώμη της πολιτικής μου ομάδας. Όπως είπε η Φαγιό επίσης, ε, επιπτώσεις αποτελεσμάτων. Το κάνει σε όλους τους τομείς η Επιτροπή, γιατί όχι στον συγκεκριμένο. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο και έπρεπε να έχει γίνει στο παρελθόν. Αν ενθυμούμε καλά, στην πρώτη συνάντηση που είχαμε για αυτό το θέμα η Επιτροπή είχε πει ότι το Frontex του είπε ότι στα αεροδρόμια αυτό θα κόστιζε σε επίπεδο χρόνου δύο δευτερόλεπτα. Ενώ στο Σαρντεγκόλ το δοκίμασαν για μία μέρα και το σταμάτησαν γιατί δεν δούλευε το σύστημα, γιατί απαιτεί το πάρα πολύ χρόνος, δεν υπήρχε αρκετό προσωπικό. Ο βαθμός ενόχλησης ήταν τεράστιος. Και ακούσαμε τι γίνεται και στο Στρασβούργο. Συνεπώς λοιπόν η μελέτη των επιπτώσεων εδώ ελείπει, οπότε θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια. Θα ήθελα να θέσω κι άλλο ένα θέμα. Γνωρίζουμε όλοι ότι σε σχέση με τις τρομοκρατικές επιθέσεις, αυτοί που διαπράττουν την επίθεση έχουν μεγαλώσει, έχουν ανατραφεί και ζουν στην Ευρώπη. Δεν είναι πρόσφυγες. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να το ξεχωρίσουμε αυτό. Σε μία από τις συναντήσεις που κάναμε, Υπόθηκε ότι, κοιτάξτε, υπάρχουν σύνορα τα οποία είναι, θα έλεγα, περίπου ανοιχτά και υπάρχει κόσμος που πηγαίνω έρχεται, ιδιαίτερα αυτοί που ζουν κοντά στα σύνορα. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά το θέμα μας είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Δεν μιλάμε για πρόσφυγες, μη συγχαίουμε τα πράγματα. Συμφωνώ επίσης και με τις ανησυχίες που ακούστηκαν για την στοχευμένη παρέμβαση και την βασισμένη σε αξιολόγηση κινδύνου. Πώς καθορίζει κανείς το επίπεδο κινδύνου. Εθνοτικό profiling. Όλους που είναι συγκεκριμένου χρώματος και οι υπόλοιποι θα περνούν. Δεν είναι ξεκάθαρο το θέμα. Να αναφερθώ επίσης και σε τρεις τροπολογίες της κυρίας Μακοβέη, την 14. Αναφέρεται ότι η προσωρινή εισαγωγή ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα στα πλαίσια των άρθρων, του άρθρου 74. Έλεγχη σύμφωνα με το άρθρο 74. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη στα εσωτερικά σύνορα μπορούν αυτόματα χωρίς να το ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσουν αυτή τη μορφή ελέγχων. Αυτό δεν πρέπει να είναι αυτόματο. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται στα εσωτερικά σύνορα αυτό το οποίο ε, ε, ε, προβλέπεται και για τα εξωτερικά στους ελέγχους, δηλαδή να υπάρχει προειδοποίηση. Τώρα, τροπολογία 21. χρήση ε, των συγκεκριμένων βάσεων δεδομένων. Γίνεται αναφορά σε ε, τρεις ε, τέτοιες βάσεις. Νομίζω ότι ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να είναι δεδομένος και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί κανείς ή αδίποτε άλλη βάση δεδομένων, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στον μικρό κατάλογο. Και τροπολογία 22. Και εδώ να πω ότι θα ήταν απαραίτητο οι βάσεις δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν λόγω των συμφωνιών με τρίτες χώρες να μην χρησιμοποιούνται αυτόματα. Να μπορούν να ελέγχονται αλλά όχι με αυτόματο τρόπο. Ευχαριστώ. Βίνμπεργκ. att vi har kontroller och jag är väldigt för de här kontrollerna och vi ser ju... Ευχαριστώ πολύ. Ε, εγώ είμαι υπέρ αυτών των ελέγχων. Διότι βλέπουμε τι συμβαίνει, βλέπουμε πόσε επιθέσει ε, λαμβάνουν χώρα, όλο και περισσότερε. Και προτιμώ προσωπικά να στέκομαι πιο πολύ ώρα στην ε, ουρά στο αεροδρόμιο περιμένοντα του ελέγχου παρά να βρίσκομαι σε πολύ χειρότερη θέση. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν καθυστερήσεις, όμως θα σκεφτούμε και την ασφάλεια. Αυτό που προτείνει η συγγήτρια είναι κάτι που καλωσορίζω. Ωστόσο, να σας υπενθυμίσω ότι οι τρομοκράτες τις περισσότερες φορές είναι ήδη ανάμεσά μας. Είναι άνθρωποι με υπηκότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή ζουν περίπου 6 έως 7.000 τρομοκράτες και δεν αρκούν οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα της Ένωρης. Πρέπει να επανεισαχθούν οι έλεγχοι και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ πιστεύω ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται και κατά την είσοδο και κατά την έξοδο. Τώρα, στην τροπολογία 18 που αναφέρεται ότι ορισμένα μέτρα θα εφαρμόζονται για μια περίοδο 6 μηνών, εγώ πιστεύω πως πρέπει να εφαρμόζονται για όσο καιρό χρειάζεται. Κύριε κυρία Μουσολίνη ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με την πρόταση γήτριας και με αυτά που είπαν και οι σκιώδεις. Είναι μια πρόταση πολύ ισορροπημένη. Ακούγοντας όμως τις συναδέλφους, τους συναδέλφους φαίνεται ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε τους σεισμούς, άρα κατασκευάζουμε επί των ηφαιστείων. Αυτή είναι η παρομή που μπορώ να κάνω. Αυτή είναι η συζήτηση που δεν λαμβάνει υπόψη το αίτημα που έχουν οι πολίτες για μεγαλύτερη ασφάλεια και η απάντηση που αυτό το κείμενο δίδεται είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν τρόπο πάρα πολύ ισορροπημένο λέει περισσότερη έλεγχη στα εξωτερικά σύνορα και να μπουν σε δίκτυο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, εντό των εσωτερικών συνόρων. Υπάρχουν τόσα συστήματα ε, που δυστυχώς δεν είναι στο δίκτυο. Αυτή είναι μια απάντηση ευρωπαϊκή η οποία επικρατεί επί των χρεοκοπημένων εγωισμών που βλέπουν να προβάλλονται σαν απαντήσεις ε, στην τρομοκρατία αυτό τον καιρό. Λοιπόν, θα θέλω να κάνω μια σύγκριση εδώ στις Βρυξέλλες όπου έχουμε το αεροδρόμιο του Ζάβεντεμ. Εμείς για να φύγουμε πρέπει ε, να πάμε τις 4 ώρες πριν στο αεροδρόμιο. Αλλά στις Βρυξέλλες, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν 6 αστυνομικές υπηρεσίες. Εάν μάλλον αν κάποιος χάσει σε μια γειτονιά το έγγραφο θα πρέπει να πάει σε αυτή τη γειτονιά γιατί μεταξύ τους δεν μιλάνε οι αστυνομικές αρχές. Ε, θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό να μην υπάρχει δικτύωση σωστή και διάλογος επικοινωνία ε, στο ε, εσωτερικό των αστυνομικών δυνάμεων. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της Βρυξέλλες. Λοιπόν, συμφωνώ με αυτή την πρόταση, δηλαδή της ενισχύσεως, αλλά πάνω απ' όλα βλέποντας ότι το γύρω και το το σύστημα του Schengen και άλλα συστήματα καλού, αναφέρονται σε διάφορες εκθέσεις που συζητούμε, θα πρέπει να υπάρχει αναμφισβήτητα τι χρειάζεται να ενισχύσουν τα εξωτερικά σύνορα και που το αναφέρουμε, αλλά δικτύωση ξεπερνώντας τους εγωισμούς των κρατών μελών όλων αυτών των συστημάτων που συλλέγουν τα στοιχεία. Πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μουσολίνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να παρέμβει. Ο κύριος Δεσόζα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που έχει δώσει προτεραιότητα σε αυτό το θέμα εξίσου σημαντική με το πακέτο για τα σύνορα του Δεκεμβρίου του 2015, την δημιουργία Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Λιμενικού. Θα ήθελα να κάνω ορισμένα γενικότερα σχόλια και μετά όταν έχουμε το κείμενο με τις τροπολογίες που προτείνεται, θα ε, τοποθετηθούμε σε συγκεκριμένες τροπολογίες. Καταρχάς, ορισμένα γενικά σχόλια. Ακούστηκε ότι η πρόταση έχει εμπνευστεί από το ζήτημα της ασφάλειας. Πράγματι. Μην βλέπετε όμως αυτή την πρόταση ως ε, ένα μεμονωμένο ε, περιστατικό. Είναι ένα μέρος μιας δέσμης μέτρων και προτάσεων που ε, έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαχειριστεί καλύτερα το μεταναστευτικό ζήτημα και τα εξωτερικά σύνορα. Αυτή Δηλαδή είναι μια πρόταση που στοχεύει περισσότερο στην ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως δεν έχει μόνο αυτό στο, στο χαστρό της. Είναι ένα μέρος του πακέτου για την μετακατάσταση, για τις νόμιμες οδούς ε, τις οποίες θα χρησιμοποιούν οι μετανάστες για να φτάνουν στην Ευρώπη. Έπειτα, κάποια μέλη της Επιτροπής σχολίασαν την έλλειψη εκτίμησης αντικτύπου και μάλιστα την έλλειψη εκτίμησης αντικτύπου σε αρκετές πρόσφατες προστάσεις της Επιτροπής. Ισχύει αυτό. Ισχύει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει συνήθως να διεξάγει εκτιμήσεις αντικτύπου. Όμως, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω πως αυτή είναι μια περισσότερο πολιτικού χαρακτήρα συζήτηση που δεν θα πρέπει να επηρεάζει το ζητούμενο εδώ. Σας διαβεβαιώ ότι αυτή η πρόταση δεν έχει γίνει ε, με άγνοια του τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Έχουμε συζητήσει με τη συνοριοφυλακή, με την ακτοφυλακή, με τα κρατημέλη. Δεν είναι λοιπόν μια τελείως τυχαία και αδικαιολόγητη πρόταση ε, ακριβώς επειδή δεν έχει γίνει εκτίμηση αντικτύπου. Και αυτό ε, πιστεύω πως είναι κάτι που πρέπει να ζητήσετε με την Επιτροπή αν έχετε τέτοιες ανησυχίες. Έπειτα, το ζήτημα της αναλογικότητας που ακούστηκε. Ε, επιτρέψτε μου να σας πω πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Τα κράτη-μέλη έχουν ήδη υποχρέωση να διεξάγουν συστηματικούς ελέγχους όλων όσοι εξέρχονται ε, της επικράτειας της Ένωσης και των πολιτών της Ένωσης. Όλοι λοιπόν που διασχίζουν τα σύνορα πρέπει να ελέγχονται. Και το γεγονός ότι ε, υπάρχει αυτός ο συστηματικός έλεγχος δεν το καθιστά θέμα αναλογικότητας. Αυτό ισχύει και σήμερα. Ο στόχος της πρότασής μας είναι κατά τη διάρκεια αυτών των συστηματικών ελέγχων να ε, γίνεται και αντιπαραβολή με βάσεις δεδομένων. Υπάρχει λοιπόν ο συστηματικός έλεγχος. Και όπως έχουμε εξηγήσει στο επεξηγηματικό σημείο αρκετά ε, ξεκάθαρα, δεν θα επηρεάσει αρνητικά τη, τα εξωτερικά σύνορα και την κίνηση εκεί. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει δώσει τη δυνατότητα για παρεκκλήσεις στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα. Ε, τώρα ποια είναι η διαφορά με αυτά τα σύνορα σε σχέση με τα, με τα εναέρια. Έχει να κάνει καταρχάς με τις υφιστάμενες υποδομές, με το πώς διεξάγεται ο έλεγχος αυτός και ε, με τη φύση των νερών. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς στο Στασβούργο και στο αεροδρόμιο που αναφέρεται, όμως ε, σε γενικές γραμμές στα, στα αεροδρόμια ο επιβάτης πρέπει να παρουσιαστεί σε κάποιο σημείο ελέγχου όπου και ελέγχεται. Και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελέγχονται με βάση την ε, υπηκότητα και την ε, ταυτότητά τους, τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα. Γίνονται λοιπόν ήδη έλεγχοι βασισμένοι σε κίνδυνο και υπάρχουν κάποιοι κοινοί δείκτες κινδύνου που χρησιμοποιούνται και που αναφέραμε εκτενώς πέρυσι ε, όταν συζητήσαμε την προσπάθεια καταπολέμησης των ξένων μαχητών, τρομοκρατών. Και στα πλαίσια της ε, μάχης κατά της τρομοκρατίας, πιστεύω πως ε, δεν είναι αυτή η πρόταση που θα είναι αποφασιστική σημασία σχετικά με την ασφάλεια. Ο στόχος είναι να πιάσουμε τους ε, ξένους τρομοκράτες μαχητές όταν προσπαθούν να βγουν ή να μπουν από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όχι να ε, ταλαιπωρούνται οι υπόλοιποι. Το σύστημα που θέλουμε να εφαρμόσουμε θα μπορεί να εντοπίσει σε ένα σημείο εξωτερικών συνόρων ενός άλλου κράτους μέλους κάποιον υπήκο άλλου κράτους μέλους που προσπαθεί να μπει. Επίσης, η δομή που έχουμε προτείνει πέρα από τους ε, υφισταμένους ελέγχους, θα προσθέσει και τους ελέγχους ε, με τις βάσεις δεδομένων. Γι' αυτό έχουμε προβλέψει αυτή τη μεταβατική περίοδο, διότι μπορεί να υπάρξει ανάγκη για επιπλέον προσωπικό, επιπλέον σημεία ελέγχου και θεωρεί το Συμβούλιο ότι έξι μήνες, τουλάχιστον η πλειοψηφία ε, του Συμβουλίου θεωρεί πως είναι ένα λογικό χρονικό διάστημα. Τώρα, εάν προταθεί ένα συντομότερο χρονικό διάστημα, είναι κάτι που θα συζητήσουμε στα πλαίσια του τρομερού διαλόγου. Τώρα, τα πράγματα είναι διαφορετικά στα χερσαία σύνορα. Εδώ, πολλές φορές εξαρτάται το πού βρίσκεσαι πώς μπαίνεις ή βγαίνεις από το χώρο του Σέγγεν, πόσοι ταξιδιώτες περνάνε τα σύνορα, πόσους συστηματικούς ελέγχους πρέπει ε, να κάνει κανείς ε, και να τους αντιπαραβάλλει με τη βάση δεδομένων. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα παρέκκλησης βασισμένη στην εκτίμηση αντικτύπου και στην εκτίμηση του κινδύνου αν αποφανθεί ότι υπάρχει κάποιος ε, συγκεκριμένος κίνδυνος σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος. Το γεγονό όμως ότι μέχρι στιγμής δεν γίνονται συστηματικοί έλεγχοι αντιπαραβαλλόμενοι με βάση δεδομένων είναι κάτι που μπορεί να θέσει κίνδυνο την ασφάλεια. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου ένα τελευταίο σχόλιο για τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, ε, δηλαδή σε περίπτωση που θα επανεισαγάγουν τα κράτη-μέλη αυτούς τους ελέγχους. Εδώ θα ήθελα να πω ότι δεν ισχύουν αυτόματα η διατάξει σε περίπτωση που ένα μέλος επανεισαγάγει ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα. Αυτή η έλεγχη, για παράδειγμα, όταν ε, γίνεται ένας αγώνας ποδοσφαίρου και θέλουν να ελέγξουν για χούλιγκαν, δεν χρειάζεται να ελέγξουν όλη τη βάση δεδομένων και όλες τις βάσεις. Δεν υπάρχει κάποιο αυτοματοποιημένο σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση οι έλεγχοι που γίνονται στα εσωτερικά σύνορα ε, γίνονται κατά περίπτωση βασισμένοι στην ανάγκη που έχει παρουσιαστεί εκείνη τη στιγμή και στην καλύτερη δυνατή ανταπόκριση. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια αυτόματη εφαρμογή όλων αυτών των διατάξεων στα εσωτερικά σύνορα της Ένωσης. Ορίστε. Αυτά κυρία Πρόεδρε είναι σε πρώτο στάδιο κάποια από τα σημεία στα οποία θέλαμε να αντιδράσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Στρέφομαι ξανά. Α, Σοφή. Πολύ σύντομα, ε. Πολύ σύντομα, λέει η κυρία Εντφέλτ. Είπε και ο συνάδελφος ότι έγιναν πολλές συνομιλίες με τους ενδιαφερομένους φορείς, εμπλεκόμενους φορείς, όπως εκπροσώπους των αεροδρομίων κλπ. Τότε γιατί δεν βλέπουμε τα αποτελέσματα των συνομιλιών. Ακόμα και δεν γίνεται ε, αξιολόγηση ε, συνεπιών για λόγους που δεν γνωρίζω, θα έπρεπε να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις ε, πληροφορίες και θα πρέπει να έχουμε και μία ανάλυση, να ξέρουμε γιατί πιστεύετε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν υποχρέωση διενεργία συστηματικών ελέγχων αντί να το εφαρμόζουν δυνητικά, να χρησιμοποιούν τις επιλογές που έχουν σήμερα για τη διενέργεια των ελέγχων. Κύριε Δεσόσα, θα θέλατε να δώσετε μια απάντηση τώρα. Στο πρώτο σημείο θα δω τι έχουμε σε κείμενο και τι μπορούμε να σας διαθέσουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Μακοβέη. Σας ευχαριστώ να πω μερικά λόγια θα ήταν καλό να δούμε κάποια από τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ακολούθησαν τις συζητήσεις με τους εκπροσώπους των μεθοριακών ελέγχων. Θέλω να πω το εξή για την έλλειψη αξιολογήσεως συνεπιών πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα και αυτό καθ' αυτό αποτελεί μελέτη αντιχτύπου Εκείνοι που διέπραξαν τις τρομοκρατικές επιθέσεις δήλθαν από τα εξωτερικά σύνορα και τα εσωτερικά. Γνωρίζουμε ότι αυτό συμβαίνει. Συνεπώς θα πρέπει να ενισχύσουμε τους μεθοριακούς ελέγχους. Τώρα μιλάμε για εξωτερικά σύνορα ως επιτοπλίστων στην έκθεση. Συμφωνώ. Θα ήταν καλό να έχουμε το υλικό που απέρευσα τις συζητήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τους εκπροσώπους των μεθοριακών ελέγχων. Αν γνωρίζουμε όμως ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτά συμβαίνουν, θα πρέπει να δράσουμε χωρίς να αναβάλουμε. Μόνο και μόνο γιατί δεν έχουμε επισήμως κάποια έκθεση συνεπειών. Κάποιοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο χάος που επεκράτησε σε κάποια αεροδρόμια όταν τα αεροδρόμια προσπάθησαν να εφαρμόσουν συστηματικούς ελέγχους. Αυτό συνέβη την πρώτη ημέρα μιας τέτοιας προσπάθειας. Καταρχάς να πω ότι όταν κάνει κανείς κάτι για πρώτη φορά μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί. Μετά όμως μαθαίνει κανείς από τα λάθη του και μπορεί η προσπάθεια να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε τα προβλήματα να μειώνονται συνεχώς για τους ε, επιβάτες. Δεν το κάνουμε αυτό για την προσωπική μας άνεση, για να μένουμε λιγότερο χρόνο στα σύνορα. Το κάνουμε για να εμποδίσουμε τους τρομοκράτες και πάνω απ' όλα να αποφύγουμε και άλλους θανάτους. Και το δικαίωμα στη ζωή είναι ε, το πρώτιστον όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια ερώτηση ίσως να μην μπορεί να απαντηθεί σήμερα αν δεν θέλετε συστηματικούς ελέγχους. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αν κάποιος λέει ότι αυτό δεν είναι καλό, δεν θέλω αυτό, τότε έχει να αντιπροτείνει κάτι. Για να είμαστε εξίσου αποτελεσματικοί ή τέλο πάντων για να δούμε ποιος εισέρχεται και ποιος εξέρχεται από τα σύνορά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μακοβέη. Όπως ήδη αναφέρατε, 28 Απριλίου στις 5 το απόγευμα είναι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροπολογίου. Ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις. Το επόμενο σημείο της ημερήσιας ε, διάταξης αφορά την πρόοδο της Τουρκίας για να πληρεί τις προϋποθέσεις για το σύστημα απελευθερώσεως από τις θεωρήσεις Πρέπει να ακολουθεί διαδικασία συναπόφαση. Γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαίρω και λεπτομερώ να μα ενημερώσει για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Τουρκία όσον αφορά τι προποθέσει για την απελευθέρωση τη απέτηση ταξιδιωτική θεώρηση. Το συζητήσαμε ήδη αυτό το θέμα, το είχαμε στη συνεδρίασή μα τη 7η Απριλίου. Όμω δεν είχαμε αρκετό χρόνο, δεν μπόρεσε να παρουσιάσει την πρόσφατη πρόοδο που σημειώθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα τη δώσω τώρα το λόγο και μετά θα ακολουθήσει συζήτηση και θα μιλήσουν τα μέλη μας. Η κυρία Σέγκατ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου και κυρίες και κύριοι. Είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετέχω στη σημερινή συζήτηση για τη δεύτερη έκθεση προόδου για την Τουρκία και τις κατά πόσο πληρεί τις προϋποθέσεις ε, για την άρση της απέτηση θεωρήσεων και έχουμε και το έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σχετικό. Δύο πράγματα να πω ευθύς εξ αρχής. Είναι σημαντικότατο να εξετάσουμε τα δύο έγγραφα που βρίσκονται επιτάπητος από κοινού. Είναι η έκθεση πρόοδου, που είναι το βασικό έγγραφο. Εξίσου σημαντικό όμως είναι να εξεταστεί και το έγγραφο εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνοδεύει την έκθεση πρόοδου αναφερόμεθα στα 72 σημεία που απαιτούνται να πληρούνται και για να ευκολύνουμε την ανάγνωση και τα επόμενα βήματα, τι κάναμε. Στην έκθεση συμπεριλάβαμε όλα όσα πρέπει να γίνουν. Οι περισσότερες πληροφορίες που σχετίζονται με τους εκπληρωθέντες στόχους εμπεριέχονται στο έγγραφο εργασίας. Α, γι' αυτό πρέπει να διαβαστούν μαζί τα έγγραφα. Δεύτερο σχόλιο αληθεύει. Την περασμένη φορά δεν είχαμε χρόνο να συζητήσουμε την έκθεση, διότι διεξήγεται πολύ σημαντική συζήτηση με τον Μάρτιν Βεβέ, τον Γενικό Διευθυντή, για τη Γενική Δήλωση για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής της Τουρκίας. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι αυτή η έκθεση πρέπει να ειδωθεί στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Ποιε είναι οι γενικέ σχέσει δηλαδή με ε, για τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία και ποια είναι η δυναμική των σχέσεων. Κυρίες και κύριοι της Επιτροπής, έχετε δει πολλά, προ... πολλά παραδείγματα διαλόγου για την απελευθέρωση από την ανάγκη θεωρήσεων. Ξέρετε ποιος είναι ο διάλογος και ποιο είναι το σχέδιο δράσης, ποιος είναι ο δικός χάρτης, ποια είναι τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, που έχουν ιστορικών και μεθοδολογία, εισαγωγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε το διάλογο με την Τουρκία για την απελευθέρωση από τις τον Δεκέμβριο 2013. Αυτό έγινε παράλληλα με την υπογραφή τη Συμφωνία Επανεισδοχή Ευρωπαϊκή Ενώσεω Τουρκία. Ο διάλογο εδράζεται επί του οδικού χάρτου. Ο οδικό χάρτη καθορίζει σαφέστατε απαιτήσει που πρέπει να πληρεί η Τουρκία για να πετύχει την απελευθέρωση από την αγκηθορήσεων. Έχουμε 72 σημεία, 72 απαιτήσει που απαριθμούνται στον χάρτη. Έχουμε πέντε κεφάλαια που σε πέντε ομάδες. Ασφάλεια εγγράφων, διαχείριση μετανάστευσης, δημόσια τάξη και ασφάλεια, θεμελιώδη δικαιώματα. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε άλλο ένα κεφάλαιο περί επανεισδοχής παρατύπων μεταναστών. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εν τω μεταξύ είχαμε δύο πολύ σημαντικές συνόδους κορυφής όπου αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έλαβαν σημαντικές αποφάσεις όσον την Τουρκία. Τον Νοέμβριο πέρσι και τον Μάρτιο φέτος. Και αυτό σημαίνει όσον αφορά τη μεθοδολογία μας και εφαρμογή για τον οδικό χάρτη σημαντικές επιταχύνσεις που απαιτούνται. Θα ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε φορά όταν μιλούμε για τα σημεία αυτά, για τις απαιτήσει. θα πρέπει να συστήσουμε βάσει της όλης καταστάσεως τι πρέπει να γίνει ούτως ώστε να πετύχουμε τον τελικό στόχο. Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε δύο εκθέσεις, την πρώτη τον Οκτώβριο του 2014 και τη δεύτερη που έχετε σήμερα εδώ μπροστά σας. Επίσης, όπως είπα εξ αρχή, γνωρίζετε ότι πρέπει όλα αυτά να ειδωθούν στα πλαίσια της γενικότερη δυναμικής των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ενώσεω με την Τουρκία. Έχουμε τις δηλώσεις συνόδου κορυφής που λέει ότι το Συμβούλιο και, Ευρωπαϊκή και το Κοινοβούλιο θα εξετάσουν το ενδεχόμενο μέχρι τον Ιούνιο φέτος να αρθούν υποχρεώσεις ταξιδιωτικών θεωρήσεων που επιβάλλουν στους πολίτες της Τουρκίας για να διέθουν τα σύνορα του Σέγγεν μόνο αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στον δικό χάρτη για τις θεωρήσεις. Θα αναφερθώ ακροθυγώ στη δεύτερη έκθεση πρόοδου, αλλά όπως ζητήθηκε και τη Σύνοδο Κορυφή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει συντομότατα την επόμενη έκθεση πρόοδου. Και σχεδιάζουμε να το κάνουμε αυτό αρχές Μαΐου, 4 Μαΐου ουσιαστικά. Λοιπόν, οι πληροφορίες που θα σας δώσουμε είναι σύντομες για να επιτρέψουμε διεξαγωγή συζητήσεως και σχόλια. Οι πληροφορίες που θα δώσω θα αναφέρονται και στις εντωμεταξύ εξελίξεις μετά τη Συνόδους Κορυφής. Έχουμε πράγματι πρόοδο, πράγματι που αναφέρθηκε και στην δεύτερη έκθεση. Οι τουρκικές αχθές προφανώς επετάχυναν την υιοθέτηση νομοθετικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσει. Στη δεύτερη έκθεση έχουμε 72 σημεία και 35 από τα σημεία τα προαπαιτούμενα έχουν καλυφθεί. Πλήρως ή σχεδόν πλήρως, μερικώς δηλαδή ανέλαβε την υποχρέωση η Τουρκία έλαβε υπόψη την αξιολόγηση των πολιτικών ηγετών και τη δική μας αξιολόγηση. Έκανε διάφορες μεταρρυθμίσεις η Τουρκία. Γίνονται πολλές αποστολές εμπειρογνωμόνων στην Τουρκία. Συνεδριάσεις επίσης μέσω βίντεο διασκέψεων και ανταλλαγής πληροφοριών μας επαφή με τους Τούρκους ομολόγους. Χρειάζεται αυτό. Έχουμε μόλις ένα δίμηνο στη διάθεσή μας. Μεταξύ δεύτερης και τρίτης εκθέσεως. Μεγάλο χρονικό διάστημα. Και εμείς και οι Τούρκοι χρησιμοποιούμε το χρόνο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να, έχουμε σαφή δεσμεύσεις από τις τουρκικές αρχές. 1η Ιουνίου να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις για την Συμφωνία Επανεισδοχής που αφορούν τους, χω... τους υπηκόους τρίτων χωρών. Έχουμε τη ρήτρα για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Η ρήτρα αυτή έπρεπε να εφαρμοστεί το 2017, μετά από ένα χρόνο. Τώρα συμφωνήθηκε επίσημα. Αυτό να εφαρμοστεί 1η Ιουνίου. Πολύ καλό αυτό. Μας βοηθάει να βλέπουμε ποια είναι τα αποτελέσματα της εφαρμογής της ρήτρα. Κυρίως τον Ιούνιο και μετά. Εξετάζουμε λεπτομερώς την πρόοδο και αξιολογούμε. Και στις πέντε κατηγορίες που ανέφερα, θα σας δώσω κάποιες λεπτομέρειες για τις πέντε κατηγορίες για να σας διευκολύνω στη μετέπειτα συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, ασφάλεια εγγράφων. Εδώ έχουμε προχωρήσει αρκετά. Έχουμε αποτελέσματα. Οι Τούρκοι έχουν ένα πολύ καλό μητρό. Αυτό είναι σημαντικό για τα εξαιρετικά έγγραφα. Οι τουρκικές αρχές χρησιμοποιούν μόνο βιομετρικά ταξιδιωτικά έγγραφα, αναγνώσιμα από μηχανήματα και συστηματικά ενημερώνουν τη βάση δεδομένων της Interpol ε, για ε, παραποιημένα και παραχαραγμένα έγγραφα. Θέλουμε να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία με τις ε, δυνάμεις της τάξης των κρατών μελών, να ενημερώνονται για τα πλαστά έγγραφα, για ταξιδιώτες που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται βελτίωση η ροή των πληροφοριών. Θα πρέπει οι τουρκικές αρχές να αρχίσουν να εκδίδουν βιομετρικά διαβατήρια που θα δίνουν στους πολίτες, στους Τούρκους πολίτες, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα δαχτυλικά αποτυπώματα των δικαιούχων. Μετά, διαχείριση μετανάστευση, στο δεύτερο κεφάλαιο. Εδώ έχουμε ένα θέμα. Καλή εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, Του σχετικού με την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Δεν είναι καινούριο σχέδιο δράση. εφαρμόζεται επί σειρά ετών μέσω εφαρμοστικών μέτρων. Είναι πολύ σημαντικό για τους όρους του οδικού χάρτη. Από τον Νοέμβριο του 2015 και πρόσφατα, μέχρι πρόσφατα έχουμε σημαντική πρόοδο. Διότι οι Τούρκοι αρχίζουν να εμποδίζουν την παράτυπη αναχώρηση, την παράτυπη αναχώρηση των μεταναστών από τις τουρκικές ακτές και να κατευθύνονται προς τις ε, ακτές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Οπότε ενισχύθηκε ο έλεγχος των Σύρων και των Ιρακινών που θέλουν να φύγουν από την Τουρκία και να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα τον Οκτώβριο είχαμε 6.000 αφήξεις την ημέρα για να δείτε πώς αλλάξαν τα πράγματα. Και τώρα έχουμε φτάσει σε λιγότερο από 200 τον τελευταίο μήνα, άρα λιγότερο από 6.000 συνολικά. Έχουμε δει πραγματική διαφορά. Άλλη σημαντική πρόοδος. Οι τουρκικές αρχές ε, έχουν εθνική νομοθεσία περί ασύλου και ειδικό φορά υπεύθυνο για τον καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα φιλοξενεί περίπου 300 ετού, εκατομμύρια ετούντες άσυλο, κυρίως Σύρους και Ρακινούς. Είναι σημαντικό να τους παρέχετε υποστήριξη και βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Παρακολούθησα τη συζήτησή σας. Ενημέρωση για την αποστολή των μελών της Επιτροπής σας στην Τουρκία. Εκφράσατε την εκτίμηση των προσπαθειών των τουρκικών αρχών που μπόρεσαν οι τουρκικές αρχές να φιλοξενήσουν τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων, να τους παράσχουν υποστήριξη. Είναι σημαντικό να το επαναλάβουμε και εδώ αυτό. Τι πρέπει να γίνει όσον αφορά τη μετανάστευση και τη διαχείριση αυτής. Οι τουρκικές αρχές θα θέσουν νέους κανόνες ε, για τις απαιτήσει για χορήγηση βίζα για πολίτες που προέρχονται από χώρες όπου υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν 11 ε, χώρες οι οποίες δεν είναι ελεύθερες θεωρήσεων για την είσοδο ε, στην Τουρκία σήμερα και η πρόταση κανονισμού η που προβλέπει κανόνες για χορήγηση αδειών εργασίας σε πρόσφυγες από άλλες χώρες εκτός Συρίας. Υπάρχει μια τέτοια πρόταση και θα ε, ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία το ταχύτερο δυνατόν. Στα πλαίσια της ε, διαχείρισης ε, της μετανάστευσης θα αναφερθώ στο θέμα της καθυστέρησης για τη χορήγηση ασύλου. 150.000 ήταν πριν μερικούς μήνες, 140.000 τώρα και υπάρχει σαφής ανάληψη υποχρέωσης από πλευράς της τουρκικής διοίκησης σε επίπεδο διοικητικό ακριβώς να επιταχυνθεί η διαδικασία και να μειωθούν οι καθυστερήσεις. Για θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας, η ε, Τουρκία έχει προχωρήσει ε, σαφώς με την ε, υπογραφή και την επικύρωση των περισσότερων συμβάσεων και πρωτοκόλων του Συμβουλίου της Ευρώπης που είχαν αναφερθεί στον οδικό χάρτη. Αναφέρομαι στη Σύμβαση και στα συνοδευτικά πρωτόκολλα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση του τράφικινγκ, για το πλήσιμο του βρώμικου χρήματος, και του πρωτόκολλο για την μεταφορά πιστώσεων. Μία ολόκληρη σειρά εμπάς περιπτώσει τα οποία είτε ήδη έχουν υπογραφεί είτε θα υπογραφούν σύντομα. Ε, η Τουρκική Βουλή έχει επίσης υιοθετήσει ένα τέτοιο νόμο που προβλέπει τη μεταφορά των συμβάσεων αυτών στην εθνική νομοθεσία της Τουρκίας. Έχουν υιοθετηθεί νομικά μέτρα πρόσφατα γύρω από τα πρωτόκολλα αυτά και παρακολουθούμε την εφαρμογή της νομοθεσίας. Δύο πράγματα πρέπει να γίνουν. Πρώτον, να επιστήσω την προσοχή σας στις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και στην υιοθέτηση του προγράμματος δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ο νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι απόλυτα ταυτόσιμος με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και είμαστε σε στιγμή επαφή με τις τουρκικές αρχές για να δούμε ποια είναι τα στοιχεία τα οποία χρήζουν βελτιώσεων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις επαφές μας και μέσω της Ευρωπόλου και την Eurojust. Ομάδα 4 τώρα, θεμελιώδη δικαιώματα. Αναφέρθηκα σε κάποιες από τις συμβάσεις προηγουμένως. Είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται. Να αναφέρω τρία στοιχεία τα οποία νομίζω είναι τα πιο ε, σημαντικά στην παρούσα φάση από τα στοιχεία του οδικού χάρτη. Το πρώτο αφορά το Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρωμά της Τουρκίας. Υπάρχει επίσης εδώ και το Εθνικό Πλάνο, η Εθνική Στρατηγική για την Επανένταξη των Τούρκων Ρωμά Παρακολουθούμε από κοντά ποια είναι τα μέτρα τα οποία προτείνονται από πλευράς τουρκικής διοίκησης και σε ποιο βαθμό εφαρμόζονται. Δεύτερον, αναθεώρηση των νομοθετικών ρυθμίσεων για την τρομοκρατία, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί με το κοινοτικό κεκτημένο αλλά και τα επίπεδα του Συμβουλίου της Ευρώπης και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τέλος την ανάγκη υιοθέτηση νόμου καταπολέμησης των διακρίσεων μέσω της δημιουργίας μιας ανεξάρτητης επιτροπής για την έρευνα πιθανών παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων από τις δυνάμεις καταστολής. Τελευταίο κεφάλαιο, επανεισδοχή, ε, ε, αναγνωρισμένη μορφής μεταναστών. Εδώ έχει υπάρξει σημαντική, επαναλαμβάνω, ο Πρόεδρος, ε, σε σχέση με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου αμοιβαίας επανεισδοχής Ελλάδας-Τουρκίας. Η Τουρκία αποφάσισε να ξεκινήσει την εφαρμογή όλων των προβλέψεων της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας από την 1η Ιουνίου θα παρακολουθήσουμε την κατάσταση προσεκτικά σχετικά με την υιοθέτηση της πλήρους συμφωνίας από τον Ιούνιο και μετά. Και η Τουρκία εφαρμόζει επίσης και τη Συμφωνία Επανεισδοχής σε σχέση με τους ίδιους πολίτες της. Εδώ παρακολουθούμε από πιο στενά την κατάσταση, το πώς λειτουργεί το τουρκικό προξενείο έτσι ώστε να εφαρμόσει πλήρως την συγκεκριμένη διαδικασία την προβλεπόμενη για την επανεισδοχή. Συμπερασματικά, είναι καιρό οι τουρκικές αρχές να κάνουν βήματα προόδου επί τη βάση συγκεκριμένων δικτών και συστάσεων που ήδη έχουν κατατεθεί στα πλαίσια της δεύτερης έκθεσης την οποία έχετε μπροστά σας. Ταυτόχρονα έχω την εντύπωση ότι μιας και η προσπάθεια συνεχίζεται με ιδιαίτερο δυναμικό τρόπο, η δεύτερη αυτή η έκθεση είναι μια έκθεση κινούμενη, εξελισσόμενη και πολύ σύντομα θα υπάρξει μια νέα έκθεση πρόοδου γιατί βρισκόμαστε στη φάση της παρακολούθησης και καταγραφής των θυμάτων προόδου σε σχέση με την δεύτερη πλέον έκθεση έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε μια καλή τρίτη έκθεση σύντομα. Θα επαναλάβω κάτι σχετικά με την απελευθέρωση του διαλόγου για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Δεν είναι η πρώτη διαδικασία την οποία έχουμε χρησιμοποιήσει και η πρώτη συζήτηση που έχουμε κάνει και μαζί σας. Ξέρετε ε, τη μεθοδολογία, ξέρετε τη σημασία για τις χώρες που εμπλέκονται, ξέρετε ότι υπάρχουν ε, πολλά ειδικά χαρακτηριστικά και ο ρυθμός εξαρτάται από την εφαρμογή η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τις εμπλεκόμενες χώρες να συνεργαστούν στενότερα με την Ένωση και να, μας, και να στηρίξουν τις δικές τους προσπάθειες ταυτόχρονα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Τουρκίας δηλαδή, στα πλαίσια της μεταναστευτικής κρίσης, μιας μόνιμης πλέον κρίσης, την οποία προσπαθούμε ε, να περιορίσουμε, να ελέγξουμε, έτσι ώστε να μην απολεστεί στο μέλλον ούτε μία ανθρώπινη ζωή στα πλαίσια των μεταναστευτικών διαδρομών. Η αποτυχία, αν θέλετε, του διαλόγου θα μπορούσε να εξηγηθεί μερικές φορές από τον επίγοντα χαρακτήρα της κρίσης. Ταυτόχρονα όμως έχουμε πλέον ένα πλαίσιο μεθοδολογικό έτσι ώστε να βοηθήσουμε να γίνουν τα πράγματα τα οποία απαιτείται. Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Αυτή ήταν η παρουσίαση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα παρακολουθήσω με ενδιαφέρον τις παρεμβάσεις των μελών της Επιτροπής σας και πιθανώς να απαντήσω και στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω αρκετούς συναδέλφους που θέλουν να παρέμβουν. Η κυρία Σπινέλη θα αρχίσει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για την όλη παρουσίαση. Επλήγηνα από τη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω την εντύπωση ότι ζω σε στον κόσμο της Καντή του Βολτέρου και έχουμε μπροστά μας τον Μακρό, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πιστεύει ότι ζει στον καλύτερο κόσμο που μπορεί να ζήσει ποτέ. Οι, ε, και οι χώρες ε, οι χώρες από τις οποίες φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι να ξεφύγουν τον κίνδυνο ονομάζονται χώρες με υψηλό κίνδυνο μετανάστευσης ευτυχώς μειώνεται ο ρυθμός αφήξεως των μεταναστών και πάνω απ' όλα έχουμε πάρα πολλές ε, σημαντικές πραγματικές εις βάθος προδιέγραψα μια σειρά επιθέτων εδώ στην Τουρκία. Υπάρχει λοιπόν ε, υπάρχουν λόγοι αισιοδοξία φαίνεται. Και απελευθέρωση των θεωρήσεων δεν συνδέεται με προόδους όσον αφορά τα, ανθρώπιν, τα δικαιώματα μάλλον, τα δημοκρατικά δικαιώματα στην Τουρκία, αλλά συνδέονται με το γεγονός ότι η Τουρκία ε, επιτρέπει το κλείσιμο των ευρωπαϊκών συνόρων, των εξωτερικών συνόρων των ευρωπαϊκών. Αυτό που ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρχει καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών, να υπάρχουν βιομετρικά διαβατήρια, να γίνεται το management της μετανάστευσης. Λοιπόν, ερωτήσεις. Πρώτη. Στη δική σας σύλληψη των πραγμάτων και ιδεών και αποφάσεων, πού και πού έρχεστε σε επαφή με την πραγματικότητα. Έρχεστε σε επαφή με τις ενώσεις, με τον ΟΗΕ, με τη Διεθνή Αμνηστία, με την Human Rights Watch που περιγράφουν αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία. Παναπατρισμό των προσφύγων προς τη Συρία, τη, τη φρικτή κατάσταση που κρατεί στους καταβλισμούς των προσφύγων στην Τουρκία, τη βία στα σύνορα με ε, την ε, Συρία, δηλαδή που πυροβολούν τους πρόσφυγες. Δεύτερη ερώτηση. Και κάτι που με εκπλήσει στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, ερώτηση. Πρέπει να συμμορφωθεί με 72 υποχρεώσεις η Τουρκία μέχρι τον Οκτώβριο του 2016. Θα πρέπει να εξαστεί νομοθεσία για την τρομοκρατία, αν θετηθεί μια νομοθεσία που λειτουργεί κατά των διακρίσεων και μεγάλο εθνικό σχέδιο για την βελτίωση της κατάστασης των Ρωμά. Πιστεύω ότι δεν θα είναι εφικτό αυτό εντός του 2016. Περιμένω μια σε έκθεση υπαριθμών 16, 17, 18 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα μας λέει ότι κινούμεθα προς τον καλύτερο δυνατόν κόσμο. Ζούμε στον καλύτερο δυνατό κόσμο. Ευχαριστώ Δεν θα επισέλθω στην ουσία αυτών των θεμάτων αυτό που παρουσιάστηκε θα πρέπει να εξετάσουμε τι λεπτομέρειε. Υπάρχει ένα ερώτημα που δημιουργείται ακολουθώντα την εκπρόσωπο τη επιτροπή Επιτροπή, ένα μέρο αυτών που είπε. Διότι μπορεί να δείχνει αυτό τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτέ, συλλαμβάνονται αυτέ οι προτάσει. Αναφέρθηκε στι συζητήσει που κάναμε χθε για την ε, επανεισδοχή στην Τουρκία. Και όλοι ήταν ικανοποιημένοι και επενούσαν τι προσπάθειε που καταβάλει η Τουρκία για τι επανεισδοχέ αλλά συνοψίζει αυτά που είπαμε λάθος. Είπαμε ότι έχει γίνει πρόοδος, αλλά η πρόοδος που έχει γίνει στον αφορά την υποδοχή των, σύρι, των Σύρων στα αντίστοιχα στο, ε, στους καταβλισμούς, αντιστοιχεί στο 11% του πληθυσμού, οι άλλοι είναι στις πόλεις και περνάνε πάρα πολύ δύσκολα οι πρόσφυγες. Και θα έπρεπε να το συζητήσουμε και αυτό. Θα ήθελα να, είμαι, να επαληθεύσω ότι δεν υπήρξε παρεξήγηση μεταξύ αυτών που λέμε εδώ και πώς αυτά ερμηνεύονται στο web stream και πώς μεταφράζονται, πώς ακούγονται μέσω της μεταδόσεως στο διαδίκτυο και πώς μεταφράζονται στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κυρία Βαλέρο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω τις εξής ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με τη Συμφωνία Επανιστοχής. Βλέπουμε ότι σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή ε, είναι τελείως ασαφή σε σχέση με τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην Τουρκία. Δεν ξέρουμε πώς έχει η κατάσταση εκεί. Ε, υπάρχουν πολλοί Τούρκοι οι οποίοι, ξέρετε, φεύγουν από την Τουρκία. Εγκαταλείπουν και η χώρα τους. Δεν είναι μόνο οι Σύριοι που εγκαταλείπουν. Όταν εγκαταλείπουν την Τουρκία άνθρωποι και γνωρίζουν ότι σε ορισμένα τμήματα της χώρας ε, τα δικαιώματα ορισμένων ομάδων ανθρώπων δεν γίνονται σεβαστά, τότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε. Ε, Ετήσεις ασύλου από το 2008 μέχρι το 2015, 72.000 αιτήματα ασύλου τότε και 150.000 αιτήματα ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοίταξα και τους υπόλοιπους πίνακες του εγγράφου και παρατήρησα ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι που ε, παραμένουν κρυμμένοι κάπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το φόβο να σταλούν πίσω στην Τουρκία. Φοβούνται την ίδια τους, για, για την ίδια τους τη ζωή. Πιστεύω πως αυτό πρέπει να το εξετάσουμε και με το θέμα των υπηκών τρίτων χωρών και των ασφαλών τρίτων χωρών. Είναι σίγουρα πάρα πολλά πράγματα που έχει επιτύχει η Τουρκία και έχει βελτιώσει το τελευταίο διάστημα. Και η Τουρκία θεωρείται ε, τρίτο, ε, ε, ασφαλές τρίτο κράτος, όμως όταν υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν από εκεί, αυτό πρέπει να μας βάζει σε σκέψεις. Από τη μία υπάρχει αυτή η συμφωνία με την Τουρκία, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε ε, τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί, προχωράμε. Και υπάρχουν κάποιες χώρες η Γαλλία και η Γερμανία μεταξύ άλλων που επιμένουν για την περαιτέρω απελευθέρωση των θεωρήσεων. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω εάν εσείς έχετε κάποιες παραπάνω πληροφορίες και τι συζητάτε ε, εκεί. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βερζιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμένα μου έχει κάνει έκπληξη το λεξιλόγιο που έχει χρησιμοποιηθεί. Ε, μου κάνει εντύπωση η ορολογία που χρησιμοποιήθηκε. Διερωτώ με πώς δουλεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή γύρω από όλα αυτά τα θέματα. Καταρχάς ε, είμαι πεπισμένη ότι δεν έχουμε με μια μόνιμη μοταναστευτική κρίση να κάνουμε, αλλά με μια κρίση προσφύγων και με μια κρίση ανθρωπιστική traite pas les Επιτροπή δεν αντιμετωπίζει τα θέματα σωστά. Και όπως είπαμε στον ΟΗΕ ότι δυστυχώς η κρίση ε, των προσφύγων θα ενισχύσει το καθεστώς αυτό το κατασταλτικό και θα οδηγήσει ε, σε ακόμα περισσότερους θανάτους στη Μεσόγειο και η επικαιρότητα δυστυχώς αυτό δείχνει με τους 400 πνιγμένους πρόσφατα. Και στην Επιτροπή μας λοιπόν συμμετέχω και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και παρακολουθώ από το 2009 που εξελέγει το θέμα της Τουρκίας με στόχο την ένταξή της ο απολογισμός τον οποίο μας κάνατε και είναι ένας απολογισμός που γίνεται τακτικά ετήσια στα πλαίσια των σχέσεων της διαδικασίας ένταξης. Υιοθετήσαμε στην τελευταία μας ολομέλεια μια έκθεση για τις σχέσεις αυτές. Η έκθεση λέει ακριβώς τα αντίθετα, μα ακριβώς τα αντίθετα σε σχέση με αυτά τα οποία εσείς μας είπατε σε πάρα πολλούς τομείς όπου η Τουρκία <clears throat> ελέγχεται. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει ουσιαστική και πραγματική πρόοδος σε σχέση με συγκεκριμένους τομείς. Αυτά τα οποία βλέπω εγώ είναι ότι οι εκθέσεις των ΜΚΙΟ, οι ε, εκθέσεις ε, της Υπηρεσίας Προσφύγων του ΟΗΕ, της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Ε, όλες αυτές οι οργανώσεις μας προειδοποιούν για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Τουρκία. Θέλετε ένα μικρό παράδειγμα. Τα σύνορα ανάμεσα στην Τουρκία και τη Συρία είναι πλέον κλειστά. Υπήρξε πριν μερικές μέρες ένα συμβάν, στα πλαίσια αυτό οι Τούρκοι συνοριοφύλακες πυροβόλησαν με πραγματικά πυρά εναντίον Σύρων και παιδιών που περνούσαν τα σύνορα. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορώ να συμμεριστώ την αισιοδοξία σας και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται την υπόθεση αυτή. Θα συμφωνήσω παράλληλα με αυτά τα οποία είπε η κυρία Γκυλιόμ. Έχω την αίσθηση ότι δεν παρακολουθήσαμε την ίδια συνεδρίαση γιατί τα στοιχεία τα οποία μας δόθηκαν, εγώ δεν ήμουν στην αποστολή για την Τουρκία, αλλά άκουσα προσεκτικά αυτά τα οποία είπαν οι συμμετέχοντες Προφανώς ε, είπαν ευχαριστούμε για την υποδοχή των τουρκικών αρχών. Γενικά όταν πηγαίνουμε στην Τουρκία και όταν μας υποδέχονται οι τουρκικές αρχές μας υποδέχονται με σωστό τρόπο. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε αυτά τα οποία μας λέγουν οι αρχές γιατί όπως υπογραμμίστηκε ήδη και από ό,τι μας λένε και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, το 90% των προσφύγων στην Τουρκία δεν ελέγχονται από την τουρκική κυβέρνηση. Θα πρέπει να το λάβετε υπόψη σας και εγώ συνεχίζω να καταδικάζω πλήρως την Συμφωνία Ένωσης Τουρκίας με τις συνέπειες. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων για τους Τούρκους πολίτες αλλά να μην επωφελούμεθα από τη συμφωνία αυτή για να μας εξηγήσετε ότι ό,τι συμβαίνει στα πλαίσια των σχέσεων Ένωσης Τουρκίας πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Δεν το πιστεύουμε αυτό και γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να διαβάσετε την έκθεση της κυρίας Πύρη που υιοθετήθηκε στην τελευταία μας οικογένεια. Επί τη βάση αυτών των νέων αξιολογήσεων θα μας δώσετε απαντήσεις διαφορετικότατες από αυτές που μας παρουσιάσατε σήμερα. Ράντα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κυρίες και κύριοι, τις ε, τελευταίες ημέρες έχουμε παρατηρήσει απειλές από μέρους της Τουρκίας. Ότι δηλαδή εάν οι Τούρκοι πολίτες δεν απολαμβάνουν ένα ε, καθεστώς απελεγμένο από υποχρεώση θεώρησης, τότε η Τουρκία θα προβεί σε αντίπεινα και δεν θα δεχτεί την επιστροφή των ε, προσφύγων. Τώρα ε, οι απειλές αυτές εντείνονται. Ο κύριος Ερντογάν είχε πει πέρυσι ότι αν θέλει θα ανοίξει τη, τα σύνορά του ε, που προς την Ελλάδα και τη Βουλγαρία και θα αφήσει τους πάντες να περάσουν. Και για αυτό το λόγο οι συζητήσεις πρέπει να συνεχιστούν μετά την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και μόνο σε αυτή την περίπτωση θα αρθεί η υποχρέωση θεώρησης. Εσείς πώς θα διασφαλίσετε ότι η Τουρκία όντως πληρεί όλες τις προϋποθέσεις χωρίς να υποκύψετε στις πιέσεις που ασκεί. Και πώς θα στηρίξετε τα κράτη-μέλη που συνορεύουν με την Τουρκία, όπως τη Βουλγαρία, εάν η Τουρκία αρνηθεί να συμμορφωθεί με αυτό το κομμάτι της συμφωνίας. Και αυξηθεί η μεταναστευτική πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μουφέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προσωπικά υποστηρίζω την απελευθέρωση των ε, θεωρήσεων για τους Τούρκους υπηκούς και για άλλες χώρες, αλλά ανησυχώ για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε το ζήτημα. Διότι όπως καταδεικνύει η συζήτηση, και η παρουσίαση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμειγνύουμε κάπως τα πράγματα. Έχουμε μια συμφωνία με την Τουρκία, μια συμφωνία που δεν μου αρέσει και πολύ και το λέω ειλικρινά για τους πρόσφυγες και έχω την εντύπωση ότι ξεπουλάμε κάπως τα πράγματα. Είπε η συνάδελφος, ε, μίλησε για τον εκβιασμό που ασκεί η τουρκική κυβέρνηση. Απελευθέρωση από τις θεωρήσεις, ναι, αλλά δεν πρέπει να χαλαρώσουμε τα κριτήρια. Θα πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια. Μιλούσαμε μακρόν για το θέμα των θεωρήσεων. Δεν καταλαβαίνω γιατί ξαφνικά όλα είναι εφικτά. Γιατί αυτό δεν ήταν δυνατό ένα χρόνο πριν, δύο χρόνια πριν, πέντε χρόνια πριν. Να έχουμε υπόψη ότι δημιουργούμε προηγούμενο εδώ διότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε διαφορετικά άλλες χώρες. Έχουμε αυστηρά κριτηρία πρέπει να πληρούνται και θα πρέπει να είμαστε εξίσου αυστηροί έναντι της Τουρκίας όπως έναντι άλλων χωρών. Δεν... Κάποιος αναφέρθηκε σε αυτά που αναφερόταν στα μέσα ενημέρωση στην Ολλανδία. Έλεγαν ότι κάποιες χώρες συμπεριλαμβανομένες της Ολλανδίας και της Γαλλίας που ήδη αναφέρονται σε προσωρινή επανεισδοχή για απαιτήσει θεωρήσεων. Ποιον ξεγελάμε, τους Τούρκους, τους πολίτες μας. Πρέπει να κινηθούμε προς την απελευθέρωση από τις απαιτήσεις θεωρήσεις σύμφωνα με τον οδικό χάρτη και ας τηρήσουμε τα κριτήρια που εφαρμόζουμε πάντοτε, διότι μόνο τότε θα είμαστε αξιόπιστοι και για τους πολίτες μας και για τους ε, Τούρκους. Ευχαριστώ κυρία Σβέμπακ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Μας είπατε ότι τα κριτήρια που πληρεί η Τουρκία είναι περίπου τα μισά από τα 72. Και μας ε, αναφέρατε επίσης ότι από το καλοκαίρι θα τεθεί σε ισχύ συμφωνία. Πώς, πώς θα διασφαλίσετε εσείς ότι η Τουρκία θα πλήρει όλες τις προϋποθέσεις. Η συμφωνία αυτή ήταν συμφωνία ανταπόδοσης. Πάρε κάποια εκατομμύρια και πάρε πίσω τους μετανάστες. Μας λέτε επίσης ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, ότι από τους 6.000 μετανάστες που έφταναν κάθε εβδομάδα τώρα έχουμε 600, όμως χθε άκουσα ότι έχουν αλλάξει οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ε, οδείωτες, ότι αυτή την εποχή πηγαίνουν από τη Λιβύη. Τι θα γίνει όμως τώρα, θα αφήσουμε να μας εκβιάσουν και εκείνοι και να τους ε, κάνουμε δώρα. Απλά μετατοπίζουμε το πρόβλημα αλλού αυτά τα πλεονεκτήματα που δίνουμε στην Τουρκία χωρίς εκείνη να πληρεί τις ε, προϋποθέσεις που πρέπει είναι απαράδεκτο. Υπάρχουν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέλη εδώ και δέκα ε, χρόνια και δεν έχουν λάβει τέτοια βοήθεια. Χρειάζεται κάποιος μηχανισμός ελέγχου για να διαπιστώσουμε αν όντως η Τουρκία πληρεί τις προϋποθέσεις και οι έλεγχοι να γίνονται τακτικά. Ευχαριστώ κύριε Λίμπερκ. Θα ζητήσω από την Ολλανδική Προεδρία του Συμβουλίου αν επιθυμεί να παρέμβει. Yes, Καλημέρα σας. Η Προεδρία εξέτασε και τα δύο αυτά έγγραφα που παρουσιάστηκαν για τον οδικό χάρτη και το έγγραφο εργασίας τον Μάρτιο του 2016 έγινε συνεδρίαση της ομάδας εργασίας. Έχουμε δήλωση για την Τουρκία του Μαρτίου του 2016 και εκεί εκφράζει τη θέση του Συμβουλίου. Ο Υπουργός Αμήνης, ο Ολλανδός, μίλησε στο Ευρωκοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα αναφερόμενος στην εφαρμογή των μέτρων. Την επόμενη εβδομάδα θα ξαναμιλήσει. Λοιπόν, επίσης το Συμβούλιο συζητεί τώρα την εφαρμογή της δηλώσεως της πρώτερης του Συμβουλίου σχετικά με την Τουρκία. Περιμένουμε την τρίτη έκθεση προόδου και βέβαια παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς όλες τις εξελίξεις και όπως είπαν και κάποιοι ευρωβουλευτές παρακολουθούμε ακριβώς τι συμβαίνει, βλέπουμε αν γίνονται σεβαστά τα κριτήρια σχετικά με τη την απελευθέρωση των θεωρήσεων και σχετικά με τη συμμόρφωση της Τουρκίας με τον οδικό χάρτη. Αυτά και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, λέει εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα σχόλια. Δεν ξέρω γιατί θεωρείτε ότι υπήρξα τόσο θετική. Ήθελα να πω ότι ήρθα να μιλήσω για το έγγραφο που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποιος είπε στην αίθουσα, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό τα έγγραφα αυτά να τα εξετάσουμε προσεκτικά και να εξεταστούν οι λεπτομέρειες. Να εξεταστεί και η έκθεση και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας. Αναφερόμαστε σε πασίγνωστη μεθοδολογία. Επί σειρά ετών ακολουθείτε. Βάση αξιολογήσεως των εργασιών μας. Αφορά 72 κριτήρια που αξιολογούνται εντός των εγγράφων. Δεν άλλαξε κάτι εν τω μεταξύ, είναι μια συνεχιζόμενη εργασία. Εγώ παρο, παρουσίασα το ιστορικό του διαλόγου για την απελευθέρωση από την απέτηση θεωρήσεων που ζητά κάποια πράγματα. Τέλος του περσινού έτους και τον Μάρτιο φέτος όλα αυτά συμπεριλήφθησαν στο γενικό πλαίσιο των σχέσεων με την Τουρκία. Δεν άλλαξε όμως η μεθοδολογία, δεν άλλαξε η προσέγγιση μας για την επίτευξη του στόχου για την απελευθέρωση από τις θεωρήσεις. Τίποτα δεν χαλάρωσε, υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται. Σας παρουσιάσαμε την πρόοδο αρχές Μαρτίου ε, και είπαμε ότι εξακολουθούμε να επεξεργαζόμεθα τα υπόλοιπα σημεία με τη συνεργασία των τουρκικών αρχών. Όπως πάντα όμως συνεργαζόμεθα με όλους τους εμπλεκομένους φορείς. Αυτή η μεθοδολογία, αυτό ήθελα να πω, είναι καλά διαθρωμένη, πολύ συστηματική. Είναι μια προσέγγιση εξέτασης διαφόρων στοιχείων, διαφορετικών, διάφορων ε, χαρακτηριστικών και δεν αμελείται τίποτα. Εξετάζουμε κάθε προϋπόθεση. Ζούμε στον ίδιο κόσμο. Ζούμε στον κόσμο της κρίσεως με άνευ προηγουμένου ροές και μια μη βιώσιμη ανθρωπιστική κρίση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι καλύτερο μπορούμε για να αλλάξουμε τα πράγματα, για να λήξει αυτή η κρίση. Ο διάλογος για την απελευθέρωση από τις θεωρήσεις είναι ένα στοιχείο, αλλά όπως είπα ευθύ εξ αρχής η μεθοδολογία προϋπήρχε και πραγματικά πειθαρχημένα εξακολουθούμε να ακολουθούμε την ίδια μεθοδολογία όπως και για τις χώρες που συζητήσατε εδώ στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Για άλλες χώρες με τις οποίες έχουμε διάλογο για την απελευθέρωση από την υποχρέωση θεωρήσεων. Θα ακολουθήσουν και άλλες. Παρακολούθησα τις συζητήσεις για την αποστολή σας στην Τουρκία και παρατήρησα μία φράση για τον αριθμό εκείνων των ανθρώπων που βρίσκονται στην Τουρκία και φιλοξενούνται. Παρακολούθησα και τα άλλα στοιχεία που θίξατε όμως, Φερρυπίν, το πώς πρέπει να πλουστεύσουμε και να διευκολύνουμε τις διαδικασίες ε, μετακατάστασης στην Τουρκία μέσω της ΥΠΑ του ΟΗΕ και να χρησιμοποιήσουμε τις μεθόδους για αυτά που γίνονται στην Ελλάδα και τα σχόλια για ενδεχόμενη χρήση ε, οικονομικών πόρων σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο. Ε, δεν άφησα τίποτα εκτός, κανένα από αυτά που συζητήσατε, διότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη δουλειά μας. Όπως είναι σημαντική και η στενή συνεργασία μας με τις ΜΚΟ και όλους εκείνους που προβαίνουν σε αξιολόγηση για την κατάσταση ε, στην Τουρκία, είτε είναι η Διεθνής Αμνηστία ή η η αρμοστία του ΙΕ για τους πρόσφυγες. Στην εισαγωγή μου αναφέρθηκα στην έκθεση που είναι πληρέστατη τόσο πλήρης και ήθελα σε κάθε κεφάλαιο να σας δώσω μία γεύση για αυτά που γίνονται. Είναι πολύ σημαντικό. Τα βιομετρικά διαβατήρια και η διαχείριση των διαβατηρίων είναι ένα από τα στοιχεία που κρίνεται. Θα κριθεί όπως κάθε άλλο στοιχείο με τον ίδιο τρόπο. Έδωσα παράδειγμα θετικών εξελίξεων, τι είχε γίνει και πριν από τις αρχές του Μαρτίου του 2016 και σας έδωσα και κάποιες άλλες πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να γίνει Πρέπει να είμαι και πρέπει να είμαι θετική, η δεμή δεν θα πίστευα στην χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία. Είναι μοναδική ευκαιρία να συνεργαστούμε με τις τουρκικές αρχές και με όλους τους άλλους τους που μπορούν να βοηθήσουν να προχωρήσουμε. Εάν εν αυτή τη ενία είμαι θετική, ναι, είμαι θετική, θέλω να είμαι θετική και αισιόδοξη, ότι αυτό θα είναι ένα από τα μέσα που θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε. Επίσης είμαι πολύ πραγματιστική. Δηλαδή ότι αυτή η μεθοδολογία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη, δομημένη καλά, έχει το ιστορικό της και είναι σημαντικότατο να εξακολουθούμε να κινούμεθα όπως παλιά για να εξασφαλίζουμε την αξιοπιστία. Για μία ακόμη φορά εξετάστε την έκθεση και το συνδευτικό έγγραφο χρειάζεται πολλή ώρα να τα διαβάσετε. Είναι μακροσκελή έγγραφο, το έγγραφο. Σας δίνει λεπτομερέστατα την εικόνα για τη συμμόρφωση με τα κριτήρια που εδώ και χρόνια ορίστηκαν στα στοιχεία του οδικού χάρτη. Αν το κάνετε αυτό, είμαστε στη διάθεσή σας να σας δώσουμε και άλλες λεπτομέρειες. Και σίγουρα θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με πολύ επικοδομητικό τρόπο συμμορφόμεν, ε, μάλλον συνεργαζόμεν, συγγνώμη, με όλους τους εταίρους και τις τουρκικές αρχές και θα σας παρουσιάσουμε μετά την επόμενη έκθεση πρόοδου που θα παρουσιάζει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, θα υποβληθεί αρχές Μαΐου και θα ξανάρθουμε εδώ ενώπιόν σας και θα συζητήσουμε. Νομίζω ότι γενικά αυτά ήθελα να δώσω σαν απάντηση, διότι νομίζω ότι αυτά που υπόθηκαν για το άσυλο και τις χώρες υποδοχής. Αυτά είναι στοιχεία που θα συζητηθούν αργότερα και οι συνάδελφοι υπεύθυνοι για το άσυλο θα σας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Σας υπόσχομαι ότι είμαστε πειθαρχημένοι και ειλικρινείς στον τρόπο που κινόμαστε στα πλαίσια του διαλόγου για την απελευθέρωση από τις θεωρήσεις. Αν θέλετε και άλλα στοιχεία για την έκθεση προόδου, είμαστε στη διάθεσή σας και στην επόμενη έκθεση θα σας δώσουμε επίσης πληροφορίες για τις πρόσφατες εξελίξεις και θα ξαναέρθουμε στην Επιτροπή για να παρουσιάσουμε την έκθεση πρόοδου και να τη συζητήσουμε μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Τιάς. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη έχει αναβληθεί μέχρι το απόγευμα τις 5.30 και θα περάσουμε τώρα στην κατοχή και απόκτηση όπλων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει επανειλημμένα συζητηθεί στην Επιτροπή μας. Υπάρχουν 245 ε, τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον εισηγητή και μετά στους Κιώδης. Η κυρία Βαλέρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Vi diskuterar eh, Λοιπόν, είναι η τρίτη φορά που συζητάμε αυτό το θέμα εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, πραγματικά. Υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις οι οποίες έχουν ακουστεί μέχρι τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί. Ο διάλογος τον οποίο είχαμε με τους υπολείπους κοιόδης ήταν ιδιαίτερα θετικός τις προηγούμενες εβδομάδες και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κάψουμε σε μια συμφωνία, να καταλήξουμε σε μια συμφωνία εκεί όπου υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ μας. Και ελπίζω να μπορέσουμε τελικά να υπερψηφίσουμε μια γνωμοδότηση την επόμενη εβδομάδα η οποία να είναι συνενετική. Ήταν δύσκολο μέχρι τώρα να ασχοληθούμε με το θέμα των όπλων. γιατί πολλοί πιστεύουν ότι δεν θα πρέπει να απαγορευθούν πλήρως τα όπλα και έχουν κατατεθεί προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Θα ήθελα να ζητήσω όμως από την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της ή να βασιστεί σε διαφορετικά κριτήρια. Είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται σε μια ιδέα αυτού του τύπου. Και εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα κάνω δικές μου προτάσεις και νομίζω ότι το ίδιο θα κάνει και η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις, η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα όπως είπα χρήσιμη και παρά τις, τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης νομίζω ότι μπορέσαμε να καταλήξουμε σε κάποιες τελικές προτάσεις θετικές. Θα ακούσω λοιπόν τις απόψεις των συναδέλφων και όλων των συναδέλφων, σκιωδών και μη, Κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να υπενθυμίσουμε και το οποίο είναι αρκετά δύσκολο ε, να συζητήσει κανείς σε εθνικό επίπεδο είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ εύκολα μια κάποια σύγχυση ανάμεσα στους κατόχους όπλων, τρομοκράτες από τη μία, κυνηγοί από την άλλη, σκοπευτές από την άλλη. Νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνονται τέτοιου είδους συγχύσεις. Οι κυνηγοί υφίστανται κρίτικες λόγω ακριβώς αυτής της ανάμιξης που γίνεται και αυτό δεν είναι σωστό. Θα ακούσω λοιπόν τις απόψεις των συναδέλφων. Uh, ο κύριος Μάλιοφ έχει το λόγο και ο δυσηγητής. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει. Πολλές τροπολογίες έχουν υποβληθεί. Και ε, η πολιτική μας ομάδα έχει υποβάλει αρκετές και καθώς και τρεις συμβιβαστικές προτάσεις. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τις δεχτεί η συγγήτρια, όμως εμείς ε, τις υποβάλαμε χάρη συμβασμού. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να υπογραμμίσω τα κυριότερα προβλήματα που είχαμε με αυτή την πρόταση, που δεν μας βοήθησαν ε, να προχωρήσουμε. Αυτή η οδηγία πιστεύω πως ε, αρχίζει ήδη με προβλήματα, διότι η τρομοκρατία που αποτελεί το πραγματικό πρόβλημα σχετίζεται με έναν νόμο που πρέπει να αλλάξει. Για να καταπολεμήσουμε την παράνομη οπλοκατοχή πρέπει να αλλάξει ένας νόμος που αφορά την νόμιμη οπλοκατοχή. Αντί όμως να κάνουμε το επιθυμητό, στοχεύουμε τους αθλητές, τους, ε, της σκοποβολής και τους κυνηγούς και επικεντρωνόμαστε στην πρόταση στην παράνομη οπλοκατοχή, στην ουσία όμως η κατοχή όπλου είναι μία από τις πιο ελεγχόμενες δραστηριότητες στην Ευρώπη. Διότι άδεια οπλοχρησίας παίρνει κάποιος μόνο μετά από ενδελεχέστα τους ελέγχους ιατρικούς και μη. Μόνο τότε μπορείς να πάρεις ε, στα χέρια σου όπλο. Και πιστεύω πως αυτή η πρόταση δεν θα λύσει το πρόβλημα ε, των όπλων που καταλήγουν στους τρομοκράτες, διότι εκείνοι θα τα προμηθευτούν από τη μαύρη αγορά. Δεν θα πάνε σε ένα νόμιμο κατάστημα, διότι φυσικά είναι και... υπάρχουν και μαύρες λίστες. Και δεν πιστεύω πως οι συλλέκτες όπλων ή οι κυνηγοί πρέπει να γίνουν ε, οι αποδιοπομπέοι τράγοι, διότι σας είπαμε, αυτόν τον τρόπο δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Και ακριβώς επειδή η πρόταση έχει ένα τόσο σημαντικό ε, πρόβλημα, θα εισαγάγει περιορισμούς οι οποίοι είναι απρόβλεπτοι. Κάτι που αναφέρθηκε στις προηγούμενες ολομέλειες και που θα ήθελα να σας πω είναι ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις μάλλον έχουν οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τέτοιες αλλαγές στην πρόταση. Οι τρομοκράτες πολλές φορές χρησιμοποιούν αυτοκίνητα για τις επιθέσεις τους. Δεν έχουμε πει όμως ότι πρέπει να αλλάξουμε τον νόμο για να εξετάζουμε και να ελέγχουμε τους οδηγούς κάθε πέντε χρόνια. Αυτό θα γίνει στην περίπτωση των κυνηγών. Δεν έχει νόημα αυτή η πρόταση. Αυτό δηλαδή είναι κάτι που δεν έχει νόημα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και ήμουν βουλευτή στην ε, Πορτογαλία και ξέρω και την ε, νομοθεσία εκεί και πρέπει να πω ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρήσουμε αυτήν την πρόταση ιδανική για την καταπολέμηση της, ε, κατα, της από τους τρομοκράτες. Δεν θα έχει κανένα απολύτω αποτέλεσμα. Το μόνο που θα επηρεάσει είναι την νόμιμη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Η οδηγία αυτή ασχολείται με την νόμιμη οπλοκατοχή. Επαναλαμβάνω και παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικεντρωθεί στην παράνομη. Αυτή η οδηγία, είπαμε, αφορά κυνηγού, συλλέκτε όπλων, αθλητές σκοποβολή και όχι στο παράνομο εμπόριο όπλων. Δεν βλέπω καμία αναφορά στο παράνομο εμπόριο όπλων εδώ στην οδηγία. Και σας παρακαλώ να μην δείξουμε προς τα έξω μία εικόνα ε, ψευδή, ότι εμείς έχουμε καταφέρει να καταπολεμήσουμε το παράνομο εμπόριο όπλων με αυτήν την οδηγία. Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν οδηγήσει σε παράνοια θα έλεγα, η οποία έχει πλήξει τους καταγεγραμμένους νόμιμους χρήστες όπλων. Ας είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη οι οποίες παράγουν όπλα, κατασκευάζουν όπλα νομίμως. οι κυνηγοί αγοράζουν όπλα που αξίζουν εκατομμύρια ευρώ. Απασχολούνται χάρη στους κυνηγού πάρα πολλοί άνθρωποι. Υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας οι οποίες θα ε, πληγούν. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κάουφμαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Οι δύο προλαλήσατε τα είπαν όλα πιστεύω. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Είναι ε, μια ατυχή σύνδεση της τρομοκρατίας με, τις, ε, με την νόμιμη οπλοκατοχή. Και πράγματι, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, πάρα πολλοί αθλητές και κυνηγοί ε, πλήττονται ακριβώς ε, από την ίδια την αιτιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρότασή της. Δηλαδή τώρα οι κυνηγοί θα θεωρούνται ύποπτοι τρομοκρατίας. Γι' αυτό θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή ακριβώς η σύνδεση να απομακρυνθεί από το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να είμαστε σαφείς και να ε, βγάλουμε το νόμιμο, την νόμιμη χρήση όπλων από αυτήν την οδηγία. Πρέπει να ενεργήσουμε με γνώμονα τη λογική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πιστεύω ότι ε, για την δική μας πολιτική ομάδα αυτό ήταν ακριβώς το κεντρικό σημείο που μας έκανε να διαφωνήσουμε κάθετα. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε διαγραφή. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα συγκεκριμένα σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη δική μας πολιτική ομάδα. Καταρχάς, τα ε, αυτόματα όπλα που αναφέρονται ε, ότι μοιάζουν με ε, όπλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πόλεμο και θέλουν, θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαγορευτούν, ότι αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κριτήριο. Υπάρχουν εμπειρογνώμονες οι οποίοι έχουν επιβεβαιώσει ότι αυτό ε, δεν ισχύει και μάλιστα αυτό μπορεί να αποβεί παραπληνητικό. Έπειτα υπάρχουν κάποια τεχνικά κριτήρια που θα έπρεπε να εισαχθούν έτσι ώστε να επιτευχθεί η ασφάλεια κτλ ποια ακριβώς είναι αυτά τα κριτήρια που θα ε, βάζουν κάποια όπλα στην απαγορευμένη κατηγορία Α. Μετά, ακούστηκαν πάρα πολλά σχετικά με τους ιατρικούς ελέγχους. Εδώ πρέπει να δούμε την προσωπική κατάσταση του ε, κάθε ανθρώπου, πώς μπορεί ε, να επηρεαστεί. Γι' αυτό πρέπει να γίνονται κατά περίπτωση εξετάσεις. Με μόνο μας εξετάσεις έτσι ώστε να μπορεί να αποφασιστεί αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος πρέπει να κατέχει όπλο ή όχι. Εγώ φοβάμαι ότι αυτό θα δημιουργήσει ένα γραφειοκρατικό τέρας από το οποίο δεν θα ξεφύγει κανείς νόμιμος κάτοχος όπλων. Χρειάζεται επίσης ε, μία ομοιογένεια κανόνων και πρέπει να ε, θεσπίζονται κανόνες και προδιαγραφές σύμφωνα με αποτελέσματα, σύμφωνα με επιστημονικά στοιχεία. Έπειτα, είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης οι αρχές που θα διεξάγουν αυτές τις, ε, αυτούς ελέγχους εμπειρογνωμοσύνης να μην ε, χρειαστεί να λογοδοτούν σε, περίπτωση, σε οποιαδήποτε περίπτωση. Μετά, θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, ασφαλή κατοχή και φύλαξη των όπλων. Στην Ευρώπη υπάρχουν ελάχιστα κοινά πρότυπα για τα όπλα και τα πυρομαχικά. Από την άλλη όμως έχουν παρατηρηθεί, το, έχει παρατηρηθεί το εξής. Ε, στο χώρο του Σέγγεν έχουν αναφερθεί μισό εκατομμύριο όπλα χαμένα που αγνοούνται, τα οποία βρίσκονται σε ε, χέρια ιδιωτών. Οι υπηρεσίες ασφαλείας της ε, Γερμανίας και ε, των κρατηδίων μας έχουν πει επίσης ότι έχουν παρατηρηθεί πάρα πολλές περιπτώσεις εγκληματικών ενεργειών ποινικών αδικημάτων από, που προέρχονται από τη χρήση όπλων από νεοναζί. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να προσέξουμε ποιοι χρησιμοποιούν αυτά τα όπλα, που δίνουμε άδειε. Επίσης, είναι, θεωρώ απαραίτητο να υπάρχει έλεγχος, επισήμανση, των σημαντικότερων στοιχείων που Ενό όπλου, από τι αποτελείται ένα όπλο. Αυτό πιστεύω θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ε, διαλεύκανση ε, εγκλημάτων. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να καταγραφούν όλες οι συλλογές από προσωπικούς συλλέκτες ή από μουσεία. Διότι, εντάξει, μπορεί να υπάρχει κάποιο ιστορικό ενδιαφέρον, κάποιο πολιτισμικό ενδιαφέρον, το οποίο να μην χρειάζεται να ελεγχθεί τόσο πολύ. Δεν χρειάζεται να καταστρέψουμε τις ιδιωτικές συλλογές που έχουν συλλεκτικό ενδιαφέρον. Επίσης, ε, δυστυχώς δεν θα μπορέσω να ακούσω την απάντηση και τη συνέχεια της συζήτησης γιατί πρέπει να προλάβω το αεροπλάνο, οπότε ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά. Σας ευχαριστώ. Ο κ. ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι συνάδελφοι υπέβαλαν 269 τροπολογίες όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άκρος ενθαρρυντικό, για δύο λόγους. Δείχνει καταρχάς ότι είναι σημαντικότατο ζήτημα για πάρα πολλούς Ευρωπαίους. Όλοι λάβαμε πολλά ηλεκτρονικά μηνύματα από οργισμένους ανθρώπους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται σε επιθετικό λόμπι όπλων στην Ευρώπη. Δεν μας γράφει το λόμπι των όπλων, αλλά οι οργισμένοι Ευρωπαίοι πολίτες όταν επιτίθεσε κατά των ανθρώπων αισθάνονται ανήσυχοι και θυμώνουν. Κάποιες τροπολογίες αντικατοπτρίζουν τη χαμηλή ποιότητα και ιδεολογική φύση της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό που είναι ενθαρρυντικό είναι ότι οι περισσότερες τροπολογίες σχετίζονται με τις ίδιες λεπτομέρειες της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πλειοψηφία πιστεύει ότι δεν υπάρχει λόγος να απαγορευθούν τα εμιαυτόματα αθλητικά όπλα ή να, να καταστραφούν ε, ιστορικά παλαιά όπλα σε ιδιωτικέ ε, συλλογές, ούτε να στιγματιστούν ομάδες ε, πολιτών και να θεωρηθούν απειλή κατά της ασφάλειας. Αυτή η Γενική Συμφωνία θα μπορούσε να αντικατοπτριστεί καλύτερα στις συμβαστικές τροπολογίες από πλευρά Θα πρέπει μαζί εμείς με την Επιτροπή ΕΜΚΟ να στείλουμε ένα σαφές σήμα προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και προς το Ευρωπαϊκό Κοινό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβλαψε πολύ την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με την πρόταση. Και δυστυχώς εμείς θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την ζημιά. Αυτό που βρίσκω κάπως ανησυχητικό βλέποντας τις ε, τροπολογίες είναι ότι πολλά από τα μέλη που σε άλλα πλαίσια τονίζουν την αναλογικότητα και την αποτελεσματικότητα και που μιλούν κατά των εκφράσεων που δημιουργούν φόβο και της χρήσεως της δημόσιας ασφαλείας ε, σαν δικαιολογία για περιορισμούς και μεγάλες αντιδράσεις, τίνουν αυτοί οι άνθρωποι να υποστηρίξουν την πρόταση, δεν υπάρχει αξιολόγηση συνεπειών. Η πρόταση συλλογικά θα τιμωρήσει 100.000 ανθρώπους που δεν έκαναν τίποτα λάθος και τίποτα κακό και θα απαγορεύσουν και θα κατασχέσουν ιδιωτική ε, περιουσία ε, και όπλα που δεν χρησιμοποιήθηκαν σε εγκλήματα για τρομοκρατία. Θα πρέπει να ε, συμμορφωθούμε με τις αρχές. Θα ήταν κάτι που εκτιμούσα. Τώρα, η διαβίβαση πληροφοριών, ε, τα πρότυπα απενεργοποίησης είναι ε, ένα πρόβλημα που πρέπει να επιληθεί και εκεί πρέπει να εστιαστούμε και όχι σε φανταστικά προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, χαίρομαι διότι κινούμεθα προς τη σωστή κατεύθυνση εδώ στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αλάχο. Δεν βλέπω άλλους από τους κοιόδης να είναι παρόντες στην αίθουσα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση. Η κυρία Ματσόλα έχει το λόγο. Thank you, Chair. Um, the original proposal... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η αρχική πρόταση συμπεριλαμβάνει τροπολογίες που στρέφονται κατά εκείνων που ασχολούνται με τα αθλητικά και κατά των συλλεκτών. Λοιπόν, μαζί με άλλους συναδέλφους έχω υποβάλει τροπολογίες για να μην υπάρξει συσχετισμός μεταξύ τρομοκρατών και των ομίμων κατόχων όπλων και δεν θα πρέπει να αναφέρονται οι πραγματικοί συλλέκτες και να θεωρούνται σαν πιθανοί ε, διευκολυντέ τη διακίνηση όπλων. Θα πρέπει να σεβόμαστε και την επικουρικότητα καλύτερα στην πρόταση, κυρίω όσον αφορά τι ιατρικέ δοκιμέ. Επιπλέον, έχουμε επαναλάβει την άποψή μα ότι οι συλλέκτε προβληματίζονται, ασχολούνται μάλλον με τι πολιτισμικέ πτυχέ των όπλων. Οι διαδικασίε επενεργοποίηση θα πρέπει να λάβουν σχετικά υπόψη την ιστορική αξία και την αναγνωρισμένη σπανιότητα κάποιων τέτοιων όπλων. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι οι τροπολογίε με αφορά το άρθρο 2 παράγραφο 2 που αναφέρεται στο ότι η οδηγία αυτή δεν θα πρέπει να ισχύει για αυτούς που είναι καλοί τυπίστοι συλλέκτες και στα μουσεία. Θέλω να έχουμε μια λογική προσέγγιση. Κοινή λογική για να αλλάξουμε την ισχύουσα νομοθεσία όταν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να κινηθούμε προς την προτινόμενη κατεύθυνση. Πιστεύω ότι τροπολογίες που επιβλήθησαν θα βελτιώσουν έτσι περαιτέρω το κείμενο που έχουν μπροστά μας και συμφωνώ με τους συναδέλφους σχετικά με αυτό. Και πραγματικά δεν πρέπει να επανεφεύρουμε τον τροχό εδώ πέρα επεξεργαζόμενοι τις τροπολογίες είδα κάποια συστήματα που ήδη υπάρχουν και σε κάποια κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσης που έχουν ισχυρό και αποτελεσματικό έλεγχο των πυροβολών όπλων. ταυτόχρονα εξακολουθούν να είναι ισορροπημένα στην προσέγγιση του. Η χώρα μου, η Μάλτα είναι ένα καλό παράδειγμα αυτού. Η νομοθεσία για τα πυροβόλα όπλα στη Μάλτα θα μπορούσε να μα βοηθήσουν να ρυθμίσουμε τι λεπτομέρειε του κειμένου όταν θα επεξεργαζόμεθα συμβιβαστικέ τροπολογίε ε, προκειμένου να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Ματσόλα. Η κυρία Γκόμε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τις ανησυχίες που εξέφρασε ο εισηγητής. Συμφωνώ επίσης και με πολλά από αυτά που αναφέρθηκαν από την κυρία Κάφμαν, την εισηγήτρια της ομάδας μου και αυτό είναι αποτέλεσμα του έργου μας σαν μέρος Επιτροπής Ασφαλείας ε, και άμυνας και που επιθυμώ να πετύχω αυτούς τους στόχους και να προωθήσω την ασφάλεια και την άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταλαβαίνοντας τη σημαντική που είναι η βιομηχανία όπλων για αυτά τα θέματα είναι βασική συνιστόσα μιας ε, βιομηχανικής βάσης για την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρώπης. Τούτου λεχθέντος εγώ είμαι υπέρ των όπλων που είναι στη διάθεση των στρατιωτικών δυνάμεων ή των δυνάμεων που ασχολούνται με την άμυνα, να περιορίσει τη χρήση σε αυτούς και να περιοριστούν όλα τα άλλα όπλα που μπορεί να είναι στην κατοχή για οδήποτε λόγο ή πρόσχημα στα χέρια άλλων. Και να μην είναι χαλαρή η έλεγχη, διότι αν δεν υπάρχουν οι έλεγχοι εύκολα μπορούν να διατίθεται τα όπλα σε μοναχικούς λύκους ή σε ομάδες που επιτίθενται κατά των πολιτών. Στη χώρα μου, αυτή την εβδομάδα, είχαμε μια συμμορία που μεταποιούσε τα όπλα των συλλεκτών, αντίκες, ό,τι θέλετε, έπαιρνε αυτά τα όπλα και τα ενεργοποιούσε. Μέσω ποινικών ε, δραστηριοτήτων, εγκληματικών δραστηριοτήτων. Τρεις μέρες μετά την επίθεση στον Πατακλάν, στο Παρίσι, η, εθνική, η δική μας η Πορτογαλική αστυνομία έκανε δημοπρασία των όπλων που υποτίθεται ήταν για συλλέκτες, για κυνηγού κλπ. Αλλά κανένας πλέον δεν τα ανοιχνεύει αυτά τα όπλα. Χρειαζόμαστε την οδηγία και δεν συμφωνώ με εκείνους που προβάλλουν διάφορα επιχειρήματα υπέρ των λόμπι των όπλων με τη δικαιολογία ότι αυτά είναι για συλλέκτες, για κυνηγού κλπ. αυτά τα όπλα. Χρειαζόμαστε αυτή την οδηγία, χρειαζόμαστε μια ισχυρή οδηγία εφαρμόσιμη που θα δεσμεύει τα κράτη-μέλη ούτως ώστε να μην συνεχιστεί αυτή η χαλαρότηση όσον αφορά τα όπλα. Σας ευχαριστώ. Η ε, κυρία Χάτ. Κυρία Χέντμαν, συγγνώμη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για μένα το θέμα της καταπολέμησης, της κατοχής και αγοράς όπλων είναι μεγάλη προτεραιότητα. Θα πρέπει να γίνεται βέβαια στα πλαίσια και στις προστασίες των προσωπικών δεδομένων και των προσωπικών ατομικών μάλλον ελευθεριών. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει σαν στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θα ήθελα η πρόταση αυτή να βελτιωθεί γιατί πολλές φορές οι προτάσεις της Επιτροπής προκαλούν αρνητικά αποτελέσματα. Υπάρχει μια μακρά παράδοση συζητήσεων στην χώρα μου γύρω από το θέμα των όπλων, ιδιαίτερα σχετικά με τους κυνηγού και τους αθλητές, σκοπευτές αθλητές. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν εμπόδια στην δραστηριότητα του κυνηγού, όπως επίσης και στις δραστηριότητες των αθλητών σκοπευτών. Βέβαια θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα για την ανιχνευσιμότητα των όπλων για να μην εξαφανίζονται τα όπλα αυτά ε, ε, στη μαύρη αγορά. Και αυτό ισχύει και για τα όπλα που έχουν στην κατοχή τους οι στρατιωτικοί. Είναι λοιπόν μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν και πρέπει να ληφθούν από όλα τα κράτη-μέλη εφόσον θέλουμε να είναι σωστά και αποτελεσματικά. Οι συζητήσεις που γίνονται ε, ε, στην Σουηδία ασχολούνται και με το θέμα των ιατρικών ελέγχων, των ιατρικών εξετάσεων. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Ε, τώρα για τα αθλητικά όπλα και τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν, τα ατυχήματα τα οποία μπορεί να υπάρξουν και τα λοιπά, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και στα πλαίσια των ιατρικών εξετάσεων. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι σωστή, απαιτείται μια πρόταση ε, καινούρια ουσιαστικά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι τα μέτρα αυτά είναι μέτρα τα οποία εκφράζουν πανικό από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν είναι σωστά μέτρα. Αν θα έλεγα παρουσιαστούν τα μέτρα αυτά μόνο και μόνο σαν μια αντίδραση στην τρομοκρατική απειλή, Αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα και στις ε, σκοπευτικές ομοσπονδίες, στις σκοπευτικές λέσχες και στα κυνηγετικά σώματα στις διάφορες χώρες, στις οργανώσεις των κυνηγών, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε ήδη πάρει πάρα πολλά mail γύρω από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη Σουηδία η συζήτηση είναι πολύ ζωηρή. Προφανώς και πρέπει να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία αλλά το 90% των όπλων τα οποία είναι θα έλεγα της μόδας, ε, στην ουσία κυκλοφορούν παράνομα, δεν ελέγχονται. Οπότε θα πρέπει να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο τα όπλα αυτά ε, φτάνουν στη Σουηδία, φτάνουν στις διάφορες χώρες. Δεν είναι μόνο το θέμα της επίσημης καταγραφής, αλλά είναι και το θέμα της εμπορίας ή λάθρα εμπορίας των όπλων που πρέπει να μας απασχολήσει. Τώρα για τα ημιαυτόματα όπλα τα οποία έχουν την όψη αυτόματων λέγεται ότι θα πρέπει να απαγορευθούν. Ε, νομίζω ότι πρόκειται για μια πρόβλεψη η οποία στερείται σοβαρότητας. Να πω επίσης ότι στην Σουηδία πάρα πολλοί λίστες ε, ε, όταν ε, εισβάλλουν σε κατοικίες για να κλέψουν χρησιμοποιούν απλά αναισθητικά σπρέι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό το οποίο έχει σημασία, λέει η κυρία Κοράτσα Μπίλτ, είναι να μην αγνοήσουμε το, την σημασία που έχει το θέμα της χρήσης και της απόκτησης των όπλων αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φοβάμαι ότι δεν έχει ε, ε, ασχοληθεί με τα πραγματικά όπλα ε, με τον τρόπο που θα έπρεπε, δηλαδή την χρήση των όπλων για άλλους λόγους και όχι για ποινικά κολάσιμες δραστηριότητες. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα τομέα ο οποίος πρέπει να μας προκαλέσει το ενδιαφέρον και να αντιμετωπίσουμε τα θέματα που δημιουργούνται. Υπάρχουν ε, πολλοί ε, πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στρέφονται εις βάρος της Ένωσης λόγω ακριβώς της σύγχυσης που προκαλείται από τα νομοθετήματα τα κοινοτικά. Ε, οι κατηγορίες των όπλων σαν παράδειγμα δημιουργούνται συγχύσεις και δεν είναι σαφείς, δεν γίνεται η διάκριση ανακατηγορία, ε, επίσης ε, σχετικά με την, χρήση, με την ονοματολογία που χρησιμοποιείται δημιουργείται παράλληλα σύγχυση. τα ημιαυτόματα είναι ββ ενώ τα αυτόματα είναι Α γενικά υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία στα πλαίσια των προτάσεων της Επιτροπής ε, δημιουργούν προβλήματα. Είναι εκτός πραγματικότητας ε, κάποιες από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απαιτούνται κοινοί κανόνες ε, και για την εξουδετέρωση των όπλων, την γιατί όταν γίνεται σωστά η εξουδετέρωση ενός όπλου δεν είναι παρά ένα κομμάτι μέταλλο, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τίποτα άλλο. Δεν θα πρέπει να μπορεί να επανενεργοποιηθεί. Και αυτό το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και δεν το κάνει η πρόταση της Επιτροπής είναι το λαφρεμπόριο όπλων. Ε, πρέπει να υπάρξουν κοινοί κανόνες και σε σχέση με τη σήμανση των όπλων ε, απαιτούνται τεχνικές ρυθμίσεις, αλλά θα πρέπει να εφαρμόσουμε καταρχάς τα ισχύοντα πρωτόκολλα και τότε θα δούμε σε ποιο βαθμό ε, χρειάζονται να λάβουμε περισσότερα μέτρα και θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα της σήμανσης του σώματος του όπλου, του σκελετού του κεντρικού του όπλου και όχι των υπολείπων στοιχείων του ε, όπλου όπως είναι ο σιγαστήρας και τα κινούμενα γενικά τμήματα. Υπάρχει επίσης και το θέμα των ιατρικών εξετάσεων στην Σουηδία. Οι γιατροί είναι αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να αναφέρουν ε, στην αστυνομία αυτούς οι οποίοι για λόγους ψυχολογικούς ή για άλλους σωματικούς λόγους δεν είναι ικανοί να κατέχουν ένα όπλο και ε, η αστυνομία ελέγχει τις άδειες κατοχής όπλων σε πενταετή βάση. Αυτό δεν βοηθάει βέβαια άλλες χώρες οι οποίες έχουν συστήματα αποτελεσματικά. Λοιπόν, απαιτείται επικουρικότητα και στον τομέα των ελέγχων. Έκδοση αδειών, ε, υποχρεωτικός χαρακτήρας έκδοσης αδειών και για την κατηγορία Β7, των όπλων Β7. Έτσι θα αποφύγουμε γραφειοκρατικές ε, περισσότερες ρυθμίσεις. Νομίζω λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν γιατί επαναλαμβάνω πολλές από τις κοινοτικέ χώρες έχουν εξαιρετικά συστήματα για τη χορήγηση αδειών και οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται με σωστό τρόπο από τις αρμόδιες αρχές. Έχουμε επίσης και ε, προβλήματα με την πώληση εξ των όπλων είναι κάτι το οποίο δημιουργεί στοιχεία ανασφάλειας. Θα πρέπει και ο πολιτής και ο αγοραστής να έχουν τα απαιτούμενα χαρτιά, τις απαιτούμενες άδειε. και αυτό πρέπει να μπορούν να το ελέγξουν οι δημόσιες αρχές. Ε, υπάρχουν πάντως ε, κάποιες μορφές πώλησης όπλων στο διαδίκτυο και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι παράνομες. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε το κείμενο και θα πρέπει επίσης ε, να ε, ε, υπάρξουν και ρυθμίσεις για την ασφαλή φύλαξη τους για την ασφάλεια για τα παιδιά σαν παράδειγμα για να μην υπάρχει κίνδυνος να πέσουν στα χέρια αυτών που θα κάνουν καταχρηστική χρήση των όπλων αυτών. Και πρέπει επίσης να υπάρξει και βελτίωση σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών, απόψεων, γνώσεων η Europol θα πρέπει να προκαλέσει περισσότερα στοιχεία συνεργασίας ε, και στα πλαίσια των ερευνών τις οποίες ε, ε, κάνουν οι διάφορες εθνικές αρχές. Ε, λοιπόν, η εναρμονισμένη ε, σήμανση των όπλων και η μεγαλύτερη συνεργασία είναι τα θετικά της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει όμως και αρνητικές πλευρές που δημιουργούν προβλήματα στους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Κυρία Κοράτσα Μπίλ, ζητήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο αν έχει να πει κάτι. Σα Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ας σχολιάσω αυτά που άκουσα. Καταρχάς να ευχαριστήσω η συγγήτρια για το σχέδιο γνωμοδότησης, το οποίο πράγματι στηρίζει πολλά σημεία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτα όμως μπω σε λεπτομέρειες. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια πάνω σε αυτά που άκουσα. Από την αρχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι η πρόταση αυτή αντιμετωπίζει θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των πολιτών εν γέννη. Δεν αναφέρεται μόνο στην τρομοκρατία. Πηγαίνει πέρα από αυτή. Εξού και οι προτάσεις που κάναμε που έγιναν μετά από ενδελεχή έρευνα και μελέτη για το που υπάρχουν κενά και ελλείψεις και προσπαθούμε με την πρότασή μας να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ελλείψεις που διαπιστώσαμε στα πλαίσια της αξιολόγησης που ε, διεξήχθη μετά από πολλούς φορείς, από εκπρόσωπους της βιομηχανίας, από ενώσεις κυνήγων, αθλητών, ε, μετά από πολλές συζητήσεις και διαβουλεύσεις που είχαμε λοιπόν με αυτούς τους φορείς σχετικά με ε, τις ε, διατάξεις της οδηγίας. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες και ε, τα παραθυράκια που έχουμε βρει, τα οποία δυστυχώς επιτρέπουν ή ε, περιέχουν τον κίνδυνο νόμιμα όπλα να μπουν στην ε, μαύρη αγορά. Αυτό που δεν θέλουμε να κάνουμε και να το επαναλάβω, να το τονίσω αυτό, είναι να κάνουμε ένα κράμα διατάξεων και να ε, κρύβεται πίσω από αυτό το ότι οι κυνηγοί εξισώνονται με τους τρομοκράτες. Είμαστε ενήμεροι για το ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες νομοταγείς πολίτες οι οποίοι ε, κυνηγούν, οι οποίοι είναι αθλητές σκοποβολής και δεν αποτελούν κανένα κίνδυνο διότι εφαρμόζουν απόλυτα τη νομοθεσία περί όπλων και οπλοκατοχής. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι εμείς δεν θέλαμε να βάλουμε ε, στο ίδιο καζάνι τους αθλητές και τους κυνηγούς με τους τρομοκράτες. Και δεν θέλαμε να περιορίσουμε την, τα δικαιώματα των πολιτών αυτών στην νόμιμη οπλοκατοχή. Επιτρέψτε μου τώρα κάποια σχόλια, τα οποία θεωρούμε αρκετά σημαντικά ε, για τα εξή θέματα. Τα, η κατηγορία Β7. Άκουσα από πολλούς ότι τα κριτήρια ομοιότητας δεν είναι σωστά κριτήρια. Και εμείς στην αρχή κιόλα είπαμε ότι γνωρίζουμε πως αυτά τα κριτήρια δεν είναι σωστά, πως χρειάζεται να δημιουργήσουμε καλύτερα κριτήρια και είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρόταση και σε οποιαδήποτε συζήτηση. Όχι μόνο στο Κοινοβούλιο, αλλά και στο Συμβούλιο. Είμαστε ανοιχτοί λοιπόν σε οποιαδήποτε πρόταση που θα μας επιτρέψει να πλαισιώσουμε καλύτερα το κείμενό μας. Τώρα, για εκείνους που το χαρακτήρισαν γελίο το κείμενό μας, να σας πω ότι από το 1991 υπάρχει αυτό το κείμενο ε, για τη συγκεκριμένη κατηγορία όπλων, τη Β1. αυτό που κάναμε είναι την ε, υποκατηγορία να την κάνουμε ξεχωριστή κατηγορία. Έπειτα, αυτό στο οποίο αποσκοπούμε και πιστεύω πως αυτή την άποψη συμμερίζεστε αρκετοί, είναι ότι δεν θέλουμε να δούμε μη αυτόματες ε, ε, εκδοχές πυροβόλων όπλων επίθεση που, που χρησιμοποιούνται ήδη από τις αστυνομικές αρχές, τις ενόπλες δυνάμεις κτλ. να πέφτουν στα χέρια αθλητών σκοποβολής. Και σίγουρα κανείς δεν θέλει να βλέπει να κυκλοφορεί νόμιμα η μη-αυτόματη εκδοχή ενός Καλάσνικοφ για σκοποβολή. Μετά κάποιος ανέφερε τα κριτήρια. Πιστεύω πως αυτό είναι μια δυνατότητα για να ε, καταστήσουμε σαφές αυτό που επιθυμούμε. Τα κριτήρια λοιπόν. Ε, τώρα, σε σχέση με τους συλλέκτες, είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την Κομισιόν. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει οδηγία, οι συλλέκτες αποκλείονται, εξαιρούνται. Και τώρα δεν θέλω να ασκήσω κριτική στους συλλέκτες, διότι σίγουρα υπάρχουν πολλοί συλλέκτες καλή πίστη, οι οποίοι είναι νομοταγείς πολίτες και ποτέ δεν έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Ωστόσο, το γεγονός ε, παραμένει ότι αυτή τη στιγμή όσα έχει οδηγία δεν έχει καμία διάταξη για τους συλλέκτες. Σύμφωνα λοιπόν με, το με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, χωρίς να αποκλείω το ότι υπάρχουν εθνικοί νόμοι που ρυθμίζουν τους συλλέκτες. Η ευρωπαϊκή λοιπόν νομοθεσία δεν περιέχει απολύτως καμία αναφορά στους συλλέκτες. Το μόνο που λέει είναι ότι η οδηγία εξαιρεί τους συλλέκτες. Πιστεύουμε πως οι συλλέκτες πρέπει να συμπεριληφθούν στην οδηγία. Το πώς θα ελέγχονται και ποιοι νόμοι θα τους διέπουν είναι κάτι άλλο. Οι βασικοί όμως κανόνες που θέλουμε να έχουμε στην Ευρώπη, που θα δημιουργήσουν με τη σειρά τους βάση για την εθνική νομοθεσία σχετικά με τα πυραβάλλα όπλα, δεν, ε, δεν περιλαμβάνουν τους ε, συλλέκτες. Συνεπώς, με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, ένας συλλέκτης έχει πρόσβαση χωρίς κανένα περιορισμό στα όπλα. Κάτι το οποίο δεν ισχύει για κανέναν άλλο νόμιμο κάτοχο όπλων αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Γι' αυτό ζητήσαμε λοιπόν να συμπεριληφθούν και οι συλλέκτες στην οδηγία. Χρειάζεται έλεγχος σε κάθε περίπτωση. Έστω να καλύπτονται από τη βασική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτά ήταν τα δύο κύρια προβλήματα που ήθελα να τονίσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Επιστρέφω στην εισηγήτρια την κυρία Βαλέρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Πιστεύω πως ε, αυτή είναι μια καλή βάση για να δημιουργηθεί μια καλή οδηγία. Ε, η γνωμοδότησή μας πιστεύω θα βοηθήσει και την Επιτροπή ΙΜΚΟ που είναι η αρμόδια Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μ' ακούτε έτσι, ναι. Επίσης να συμφωνήσω και εγώ με πολλά από τα οποία υπόθηκαν. Ε, η εικόνα που έχουμε δημιουργήσει με αυτή την πρόταση στους ε, αθλητές, σκοποβολείς και στους κυνηγούς είναι όντως άσχημη. Και σίγουρα δεν έχουμε αποκτήσει την καλύτερη φήμη όσοι, εμείς, όσοι ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα. Αυτό το φαίνεται και από τις πολλές τροπολογίες που υποβλήθηκαν. Σίγουρα αυτή η συζήτηση είναι ιδιαίτερη Και μου κάνει εντύπωση πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ε, λέει τώρα πως ε, δεν είναι αυτή η πρόθεση που είχαμε και τα λοιπά να βάλουμε ε, στο ίδιο καζάνι τους αθλητές και τους κυνηγούς με τους τρομοκράτες. Ακούσαμε τις απόψεις ε, και πολλών πολιτικών ομάδων και πολλών ε, κρατών μελών. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει διαφορετική εθνική νομοθεσία. Γνωρίζουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι στην Ισπανία οι κανόνες είναι πολύ πιο χαλαροί, η νομοθεσία μάλλον πολύ πιο χαλαρή από ό,τι στις σκανδιναβικές χώρες για την όπλοκατοχή και για την έκδοση άδεια για όπλο. Σίγουρα πρέπει να προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε την νομοθεσία εκεί όμως χρειάζονται γι' αυτό κάποια βασικά κριτήρια τα οποία θα πρέπει να ισχύουν για όλους. Για παράδειγμα, ιατρικές εξετάσεις που θα επιτρέπουν ε, στον ε, χρηστή την, ε, να λάβει άδεια για όπλο. Φυσικά δεν μπορούν να αποκλειστούν τα λάθη από κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύω πως μπορούμε να βοηθηθούμε με τη... και να ακολουθήσουμε βέλτιστες πρακτικές για να βρούμε το καλύτερο δυνατό ε, τρόπο. Σίγουρα κάποιο πιστοποιητικό από γιατρό θα βοηθούσε. Ε, θα ήθελα τώρα να πω ότι ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις εισηγητές και τους ευχαριστώ και για τις οπτικές γωνίες που έδωσαν από τα δικά τους κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις πανεμβάσεις, συνάδελφοι. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ανακοίνωση για ισχυρότερα και πιο ευφυή συστήματα πληροφορική για την ασφάλεια των συνόρων. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανακοίνωση αυτή και μετά θα δώσω το λόγο στα μέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τον κύριο Σλόν από την DG Home. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά την ανακοίνωση για πιο ισχυρά και πιο ευφυή συστήματα πληροφοριών για την ασφάλεια των συνόρων, είναι σημαντικό αυτό για αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 100 μελών για τη διαχείριση των συνόρων και την επιβολή ε, του νόμου. Αυτό ήταν κάτι αυταποδείκτο. Τονίστηκε και στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια και στα διάφορα διαδοχικά συμπεράσματα των συμβολίων. Επί σειρά ετών οι ανάγκες εκαλύφθηκαν από συστήματα που αναπτύχθηκαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώση και μελών και έτσι οι μεθοριοφύλακε, οι αστυνομικοί και οι διάφορε αρμόδιε αρχέ έχουν τι αναγκαίε πληροφορίε για άτομα σύμφωνα με του σκοπού και τη λειτουργία του κάθε φορέα. Τώρα πρέπει να πάμε στην επόμενη φάση. Δηλαδή να δούμε πώς αυτά τα συστήματα που εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς μπορούν να γίνουν αποτελεσματικότερα. Ποια νέα συστήματα πρέπει να αναπτυχθούν και πώ η αρχιτεκτονική δομή διαχείριση των στοιχείων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να ενισχυθεί. Και αυτό είναι ο σκοπός της ε, ανακοίνωση. Η ανακοίνωση αναφέρει το SIS, το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν, το Eurodac και το σύστημα ε, για τις θεωρήσεις, το PRUM, το API, το Europol, το ECRIS το τελωνιακό σύστημα και τη βάση δεδομένων της ε, Europol. Εν γέννη, αυτά τα συστήματα πληροφοριών παράγουν χρήσιμα αποτελέσματα και κάποια από τα συστήματα λειτουργούν πολύ καλά. Όμως η ανακοίνωση εντοπίζει και σειρά ελλείψεων όπως η υποβέλτιστη λειτουργία των παρόντων συστημάτων και να όσον αφορά τις πληροφορίες που δεν καλύπτουν κανένα από τα υπάρχοντα συστήματα και υπάρχει ένα περίπλοκο τοπίο ε, συστημάτων που τα διαχειριζόμαστε με διαφορετικό τρόπο. Ε, ας αναφερθώ σε κάποια από τα κενά. Το σύστημα πληροφοριών Schengen είναι το μεγαλύτερο και το πιο χρησιμοποιούμενο σύστημα για τη διαχείριση των συνόρων και για τις δυνάμεις τάξης εμπεριέχει πάνω από 63 εκατομμύρια ε, σημεία συναγερμών, αν θέλετε, ε, ε, έχει χτυπήματα χρησιμοποιήθηκε από 2 εκατομμύρια τελικούς χρήστες. Όμως σημαντική λειτουργία λείπει σήμερα από αυτό. Αν πρέπει να ψάξεις ένα όνομα στο σύστημα, μπορεί να το ψάξεις το μέσο ονόματος, αλλά όχι βάσει δαχτυλικών αποτυπωμάτων να γίνει έρευνα. Δηλαδή δεν υπάρχει συναγερμό στο SIS, ε, κάποιο όμω που καταστείται το SIS και χρησιμοποιεί ένα ε, πλαστό έγγραφο μπορεί να ξεφύγει. Η ανακοίνωση αναφέρεται ότι χρειάζεται αυτό με το σύστημα δαχτυλικών αποτυπωμάτων όπως το ΕΦΙΣ και θα πρέπει να αναπτυχθεί ε, και έχει μέγιστη προτεραιότητα να μπορεί να αναγνωρίζει και να αναζητά βάσει δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Δεν καλύπτονται όλες οι ανάγκες για πληροφορίες από τα εφιστάμενα συστήματα. Χρειάζεται ένα σύστημα για υπηκόστη των χωρών, για είσοδο-έξοδο. Ε, παραμένουν όμως άλλα κενά. Αναφερόμαστε στην ανακοίνωση υπήκοοι των χωρών που εξαιρούνται από θεωρήσεις και δεν υπάρχουν στοιχεία API, για αυτούς τους ταξιδιώτες δεν υπάρχουν ε, πληροφορίες πριν καταφτάσουν αυτοί οι άνθρωποι σε εξωτερικά σύνορα Σέγγεν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν το τέλος του έτους θα διερευνήσει κατά πόσο είναι δυνατόν τεχνικός και κατά πόσο θα ήταν αναλογικό να υπάρχει ένα σύστημα εγκρίσεων ε, και ταξιδίων για αυτού του ταξιδιώτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Τώρα το ότι δεν είναι συντονισμένα τα συστήματα και δεν επικοινωνούν. Οι διάφοροι φορεί αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πρόσβαση πολλαπλών συστημάτων που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα κράτη-μέλη δεν συνδέονται με όλα τα συστήματα που υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω. και αποθηκεύεται διαφορετικά η πληροφορία σε διάφορα συστήματα που δεν είναι συνδεδεμένα. Η ανακοίνωση εντοπίζει λοιπόν τέσσερις στόχους για καλύφθουν τα προβλήματα. Για να κινηθούμε προς πιο ευφυή και ισχυρά συστήματα όσον αφορά την προστασία των σύνορων. Πρώτος στόχος. Αυτό το σύστημα πληροφοριών θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό, επικαλύψεις πρέπει να αποφευχθούν και οι φυστάμενες επικαλύψεις να εξαλειφθούν και να θα πρέπει να καλυφθούν και να αντιμετωπιστούν. Θα πρέπει να ακολουθηθεί προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τη εξελίξη τεχνολογικής και θα πρέπει εξ σχεδιασμού να προστατεύεται ιδιωτική ε, ζωή. Τρίτον, πρέπει να γίνουν σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των τρίτων χωρών. Απ' την αρχή θα πρέπει να προστατεύονται ε, εφαρμόζοντα τη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τέταρτον, όπου είναι αναγκαίο και εφικτό, τα συστήματα πληροφοριών θα πρέπει να διασυνδέονται και να προβλέπεται διαλειτουργικότητα. Ταυτόχρονα, ταυτόχρονη έρευνα των συστημάτων θα πρέπει να εξασφαλίζεται. Να συλλέγονται όλες οι πληροφορίες για τους μεθοριοφύλακε και για του αστυνομικού. Όταν και όποτε χρειάζεται αυτό για να εκτελέσουν το καθήκοντά τους. Σύμφωνα με την ενδεδειγμένη πρόσβαση σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της προστασίας των δεδομένων για να τονωθεί αυτή η διαδικασία προ τη λειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει μια ομάδα εμπειρογνωμών ψηλού επίπεδου με, με διάφορους φορείς, εθνικούς φορείς, διεθνείς φορείς, εμπειρογνώμων κλπ. θα συμμετέχουν. Η πρώτη συνεδρίαση τη εν λόγω ομάδα προβλέπεται να γίνει στα μέσα Ιουνίου. Η ομάδα θα εξετάσει νομικά, τεχνικά και επιχειρησιακά προβλήματα για να πετύχουμε τη διαλειτουργικότητα που θέλουμε των συστημάτων και καθώς να εξετάσει την αναγκαιότητα, την αλογικότητα και τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα εφιστάμενα συστήματα και τι θα γίνει με τα στοιχεία. Θα αναπτύξει στατικικό όραμα για διαλειτουργικότητα με συγκεκριμένες δράσεις βράχη πρόθεσμα, μέσο πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Εν τω μεταξύ δεν θα σταματήσουμε τις προσπάθειες. Αντιθέτως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μια σειρά συγκεκριμένων δράσεων. Πολλές από αυτές τις δράσεις θα λάβουν χώρα το 2016. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύντομα θα υποβάλει πρόταση προς αναθεώρηση της νομικής βάσης του Eurodac, ούτως ώστε να διευρύνουμε περαιτέρω τη λειτουργικότητα αυτού όσον αφορά ε, την, ε, τους ε, παράτυπους μετανάστες στην επιστροφή αυτών. Θα προτείνουμε αναθεωρημένη νομική βάση για το SIS, ε, το σύστημα πληροφοριών του Σέγγεν, μέχρι το τέλος ενεστώτος έτους και θα εξετάσουμε τη δυνατότητα για περαιτέρω βελτιώσεις για το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις. Θα αξιολογήσουμε την ανάγκη να αναθεωρήσουμε τη νομική βάση για την επεξεργασία των στοιχείων API. Θα παρουσιάσουμε τους επόμενους μήνες και μέτρα για την ασφάλεια των εγγράφων και τη διαχείριση των ταυτοτήτων και να ενισχύσουμε την καταπολέμηση κατά των, της παραποίησης των εγγράφων. Θα υποβάλουμε σχέδια αποφάσεις για τεχνικές επιδόσεις αργότερα για την ανάπτυξη του ΕΦΙΣ και όπως αναπτύχθηκε θα καλύψουμε και την ανάγκη, θα δούμε αν δυνατόν να έχουμε ένα σύστημα που θα δίνει πληροφορίες για τις μετακινήσεις στα ταξίδια και χορήγηση αδειών. Τώρα για τη διαλειτουργικότητα θα συνεργαστούμε με την UNISA, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία που διαχειρίζεται ε, τα διάφορα συστήματα. Θα εξετάσουμε τα σημεία διαπαφής για την έρευνα, πώς θα μπορεί να γίνει ταυτόχρονη έρευνα σε πολλά ε, συστήματα ταυτόχρονα χωρίς να επηρεαστούν τα εφιστάμενα δικαιώματα πρόσβασης. Η UNISA και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δει ποια είναι η διατηρικότητα μεταξύ κεντρικών συστημάτων, αν μπορεί να προωθηθεί η διατηρικότητα των συστημάτων πέρα από τη διασυνδυσιμότητα που προβλέπεται μεταξύ του συστήματος για τις θεωρήσεις και του συστήματος που εξετάζει εισόδους-εξόδους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε αν είναι δυνατόν να υπάρχει και σύστημα διαχείρισης των βιομετρικών στοιχείων και όλα τα συστήματα που χρησιμοποιήσουν από κοινού τα βιομετρικά στοιχεία και κατά πόσο μακροπρόθεσμα μπορεί να αναπτυχθεί ένα κοινή, μια κοινή βάση δεδομένων, κοινή αποθήκη του επίνεντος εισαγωγικών δεδομένων. Μαζί με την Ελίσσα θα προχωρήσουμε προς ομοιόμορφη ε, μορφή έρευνας για τα συστήματα πληροφοριών. Θα εξετάσουμε κατά πόσο μπορούμε να συμπληρώσουμε και το σύστημα Europol για την έλευνα, για τους εγκληματίες κλπ. Πιο γενικά. Η Λίζα θα, η θα έχει δυνατότητα να ελέγχει και την ποιότητα των στοιχείων που εξετάζονται, ε, που χρησιμοποιούνται από όλα τα συστήματα που ελέγχει. Θα πρέπει να προωθήσουμε τη χρήση των συστημάτων των κάτι μέλη. Ζητούμε τα κάτι μέλη να μεγιστοποιήσουν τη χρήση του SIS, εισάγοντας σχετικές πληροφορίες και συμβουλευόμενα το σύστημα όποτε αυτό απαιτείται. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ηλεκτρονική διασύνδεση με τα εργαλεία της ε, Europol σε όλες τις, τα σημεία διαλέψης εξωτερικών συνόρων. Θα συνεργαστούμε με την Europol να προωθήσουμε συνεργασίες μεταξύ του συστήματος πληροφοριών της Europol με άλλα συστήματα, κυρίως το σύστημα πληροφοριών ε, Schengen. Εν κατακλείδη, αυτό το θεματολόγιο είναι φιλόδοξο. Απαιτείται συντονισμένη δράση. Η ανακοίνωση δεν προσφέρει μια γρήγορη λύση. Θα χρειαστούν χρόνια να εφαρμοστούν όλες οι προτάσεις και να καταλήξουμε στα σωστά επίπεδα. Δηλαδή η αρχιτεκτονική δομή για τα σύνορα και την ασφάλεια θα είναι πλήρε σύστημα, θα υπάρχει πλήρη διαλειτουργικότητα και όλα θα λειτουργούν όπως πρέπει. Αυτό πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς και προϋποθέσεις εδώ με Εφαρμογή και υλοποίηση της ανακοινώσεως είναι δύσκολη, αλλά είναι αναγκαία για να προστατεύσουμε καλύτερα εξωτερικά σύνορα και για να βελτιώσουμε την εσωτερική μας ασφάλεια και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ποιος? Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση. Βλέπω με ικανοποίηση ότι μας δείχνουν με συνολικό τρόπο την κατάσταση, πού βρίσκονται τα προβλήματα και ποια είναι τα νέα βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν με προγραμματισμένο όμως τρόπο. Ξεκινώντας θα ήθελα να αναφερθώ στο σύστημα πληροφοριών Schengen παρά τα πολλά προβλήματα σε επίπεδο προϋπολογισμού, νομίζω ότι το σύστημα αυτό ενημέρωσης χρησιμοποιείται με σωστό τρόπο. Βρίσκεται ήδη στη δεύτερη φάση εφαρμογής και με την εισαγωγή του συστήματος ψηφιακών αποτυπωμάτων και αυτό θα έλεγα θα μας επιτρέψει να κάνουμε περισσότερες βελτιώσεις από ό,τι μέχρι τώρα. Και σχετικά με το SIS και τη διαδικασία γύρω από το SIS, το Κοινοβούλιο έχει υπερασπιστεί το μέσο αυτό. Αντίθετα από πάρα πολλά κράτη-μέλη δεν ήταν ιδιαίτερα θερμά με την πρόταση αυτή αλλά νομίζω ότι το σύστημα τελικά επικράτησε. Για μια ακόμη φορά λοιπόν είμαστε σε θέση να προγραμματίσουμε σωστά τα μελλοντικά μέτρα και νομίζω ότι οι αποφάσεις για τις επαναπροωθήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο SIS. Έχω αρκετές ερωτήσεις να θέσω. Καταρχάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι είναι χρήσιμο να ανακοινώσει ότι κάποιες νέες προτάσεις ε, ε, θα κατατεθούν σύντομα όταν παράλληλα δημιουργείται μια ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία θα εξετάσει ε, ε, τις πιθανές επικαλύψεις στα συστήματα που χρησιμοποιούνται. Δεύτερον, σήμερα έχουμε μια υπηρεσία για τη διαχείριση των πληροφοριών και δεν ε, μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό. Απαιτείται να υπάρχει ε, η εντολή η οποία θα επιτρέψει στο σύστημα να προσαρμοστεί στις ανάγκες που μπορεί να αλλάζουν. Τρίτον, ε, σχετικά με τους λογιστικούς ελέγχους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως πρέπει να αναθεωρήσει το, την νομική βάση για το Eurodac. Αυτό μπορεί να το κάνει ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα μέτρα που έχει στη διάθεσή της και πώς θα χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Eurodac για να παρακολουθεί τις λεγόμενες κινήσεις δευτέρου επίπεδου ή δευτερεύουσες κινήσεις. Ε, πέμπτον, η ποιότητα της πληροφόρησης θεωρείται ένα οριζόντιο πρόβλημα από την Επιτροπή και ε, απαιτεί την δημιουργία μιας κεντρικής ικανότητας αξιολόγησης της ποιότητας των δεδομένων. Δεν το καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Και μια τελική, ε, τελευταία μάλλον ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν νέα μέτρα για τα, έγγραφα, για τα ηλεκτρονικά έγγραφα και την ασφάλειά τους. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τι ακριβώς θέλει να κάνει γύρω από το θέμα των ηλεκτρονικών εγγράφων. Ευχαριστώ κύριε Κοέλιο, η κυρία Φαγιό. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Χαιρετίζω τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποβάλει προτάσεις και ένα σχέδιο δράσης σχετικά με το πώς στο μέλλον θα χειριζόμαστε με τον κατάλληλο τρόπο τα δεδομένα. Όπως είπε και ο κύριος Κοέλιο, θα ήθελα και εγώ να θίξω ορισμένα σημεία και να κάνω κάποιες ερωτήσεις, διότι ε, επικρατεί μια σύγχυση. Βλέπει η Επιτροπή ένα μελλοντικό ε, μια μελλοντική κεντρική βάση δεδομένων. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε. Έχουμε την ε, βάση δεδομένων PNR με τα δεδομένα των επιβατών, τη βάση Schengen, πολλές βάσεις δεδομένων τις οποίες χρησιμοποιούμε και αναρωτιέμαι εάν αυτό το σχέδιο δράσης συμφωνεί με όλα αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε μέχρι τώρα για τα ευφύ σύνορα δηλαδή και για άλλα σημαντικά θέματα. Πώς το πρόσφατα έγκριθεν πακέτο για τα προσωπικά δεδομένα θα καταφέρει να ενώσει διαφορετικές κατηγορίες επιβατών, ταξιδιωτών, δηλαδή ταξιδιώτες, πρόσφυγες, μετανάστες, ε, ταξιδιώτες με θεώρηση, χωρίς θεώρηση και έγινε και μια πολύ καλή ερώτηση σχετικά με τους εμπειρογνώμονες. Εκείνοι θα εξετάσουν παράλληλα διάφορες άλλες εναλλακτικές επιλογές. Θα μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα επηρεάσει η πρόταση αυτή το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Φαγιόν. Η κυρία Μίλναρ, σας ευχαριστώ. Και εγώ θα κάνω ερωτήση παρόμοια με εκείνη των ε, συναδέλφων. Καταρχάς να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθε να συζητήσει το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας. Όπως γνωρίζετε όλοι θέλουμε να προστατεύσουμε το Σέγγεν από την κατάρρευση και να δημιουργήσουμε κάτι καλύτερο, κάτι καινούριο. Η έλεγχη όμως στα σύνορα δεν είναι λύση. Έχω Κάποια σχόλια όμω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει τη δημιουργία ενό κεντρικού συστήματο εισόδου και εξόδου. Και όπω είπε και η κυρία Φαγιών, και εγώ θεωρώ ότι δεν μας λείπουν τα δεδομένα. Το πρόβλημα είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση και η διαλειτουργικότητα. Επίσης υπάρχει έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη για την επεξεργασία των δεδομένων. Γι' αυτό λοιπόν θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ε, πει παραπάνω πληροφορίες για το σύστημα το οποίο δημιουργούν και να μας πείσει για τα ωφέλη που θα έχουμε στον τομέα της ασφάλειας. Έπειτα, η διατήρηση δεδομένων και οι περιορισμοί. Η απόφαση του δικαστηρίου ε, μας καθιστά δύσκολο να δημιουργήσουμε μία περίοδο διατήρησης δεδομένων που θα βοηθήσει στην αύξηση της ασφάλειας. Επίσης, τα βιομετρικά δεδομένα θα έχουν και θετικές και αρνητικές επιπτώσεις. Ποιες ε, ασφαλιστικές δικλείδες προβλέπονται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη και χρήση μετά των δεδομένων αυτών. Έπειτα, η ανακοίνωση εστιάζει στην παράτυπη μετανάστευση και όχι στον ε, εξυγχρονισμό των ε, συνόρων που θα οδηγήσει και στην αποτελεσματικότερη ε, φύλαξή τους. Καταλαβαίνω το σκεπτικό, όμως η πρόκληση δεν θα έπρεπε να είναι να αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα ταυτόχρονα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άλμπρεχτ, ευχαριστώ και εγώ για την παρουσίαση. Συμφωνούμε, πιστεύω όλοι, ότι η καλύτερη πρόσβαση στις ε, πληροφορίες που διαθέτουμε και η καλύτερη διαχείρισή τους είναι αυτό που χρειαζόμαστε για να εντοπίσουμε ύποπτε δραστηριότητες. Επίσης, σχετικά με την ε, διαχείριση των συνόρων και με την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, να πω πως ε, χρειάζεται να μην ξεχνάμε τι διακυβεύεται εδώ. Επίσης, ως προς τη διαλειτουργικότητα. Χρειάζεται διαλειτουργικότητα για να διευκολυνθεί και η πρόσβαση στην πληροφορία. Όμως το θέμα εδώ δεν είναι μόνο θεωρητικό. Όταν μιλάμε για πρότυπα πρέπει να δούμε στην πράξη τι θα γίνει. Ας δούμε για παράδειγμα το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν, τη Eurodac, το σύστημα για τις θεωρήσεις, την Ευρωπόλ, ε, όλες αυτές τις βάσεις δεδομένων, το πρόσφατο PNR και άλλε βάσεις ε, δεδομένων και ας δούμε τι συμβαίνει με την προστασία δεδομένων. Θα παρατηρήσετε ότι υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα για κάθε διαφορετική βάση δεδομένων. Καταφέραμε στα πλαίσια τη αστυνομική συνεργασία να ε, επιτύχουμε μία ασφαλή επεξεργασία και φύλαξη δεδομένων. Και αυτό χάρη στη δουλειά όλων μας. Όμως αυτή η οδηγία δεν, δεν θα ισχύει στα συστήματα που αναφέρατε. Αν θέλουμε να επιτύχουμε αυτήν την συνοχή και αν θέλουμε πράγματι να ενοποιήσουμε τα ε, στάνταρτ, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτείνει ενιαία πρότυπα για όλους. Δεν καταλαβαίνω. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχει ζητήσει επανειλημμένα. Θέλουμε ε, ομοιόμορφα πρότυπα στην προστασία δεδομένων. Εντάξει, τα κράτη-μέλη έχουν τα δικά του συστήματα, ωραία. Τι θα γίνει όμως με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες πώς θα επιτύχουμε αυτήν την ομοιογένεια εκεί. Πρέπει να ακολουθούμε και εμείς τα πρότυπα που επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη και να τα εφαρμόσουμε αμέσως στα διαλειτουργικά συστήματα και στις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων. Επίσης, όπως είπε και η συνάδελφος νωρίτερα, να αναφερθούμε και στους περιορισμούς που έχουμε, που πρέπει να εφαρμόσουμε και να υπερπηδήσουμε πολλές φορές. Γι' αυτό χρειάζεται περισσότερη πληροφόρηση. Χρειάζεται να τοποθετηθεί το δικαστήριο για την ε, χρονική περίοδο διατήρησης των δεδομένων, για τους περιορισμούς που πρέπει να υπάρχουν και μετά ε, θεωρώ επίσης ότι πρέπει να είμαστε σαφέστατοι σχετικά με το τι θέλουμε, με τις διαφορετικές περίοδους διατήρησης των δεδομένων, με τους περιορισμούς ως, πως, ως προς τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, για τις κατηγορίες δεδομένων και για τη μέγιστη χρονική περίοδο διατήρησης. Εδώ θα ήθελα μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση όχι απλά να λέμε ότι όλα αυτά τα συστήματα είναι διαλειτουργικά, αλλά το καθένα έχει τους δικούς του κανόνες. Χρειάζεται συνοχή. Ευχαριστώ κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν είχα ζητήσει το λόγο. Αλλά εφόσον είμαι σκιώδης, θεώρησα ότι ήταν φυσικό Καταρχάς να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω ένα έγγραφο που παρουσιάζει όλα τα συστήματα επεξεργασίας των δεδομένων. Διερωτώ με αν ακολουθούμε σωστή προσέγγιση. Τώρα, πολλές αναθεωρήσεις γίνονται παραλλήλως Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα σύστημα άλλο που θα δημιουργήσουμε στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας, όπως και ο κύριος Άλμπρεχτ. Θέλω εναρμονισμένο. Εναρμόνιση εν συγκρίση με τι. Η διαλειτουργικότητα με τρομάζει. Ποιοι είναι οι στόχοι. Διότι τελικά καλύπτουμε πολλά διαφορετικά πράγματα που πρέπει να είναι διαλειτουργικά με διαφορετικούς στόχους. Ετούντες άσυλο, κλεμμένα έγγραφα ε, σε σημασμένα άτομα από την Europol κλπ. Θα αυξηθούν τα στοιχεία. Είπατε μόνο για το σύστημα SIS 3 δισεκατομμύρια χτυπήματα αναζητήσεις. Τι κάνουν με όλη αυτή την πρόσβαση. Αυτό είναι το ερωτηματικό που έχω πάντα. Τα τεχνικά εργαλεία, τα τεχνολογικά εργαλεία δεν λύνουν τα πάντα και δεν θα επιλύσουν ποτέ τα πάντα. Εγώ φοβάμαι όταν δημιουργούμε όλα αυτά τα συστήματα και ξέρουμε ότι κάτι μέλη μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν άσχημα, όπως και το ΣΥΣ κύριε Κοέλιο. Έχω κάποιες πληροφορίε για τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί στη Γαλλία. Μου δημιουργεί ερωτηματικά πώς λειτουργεί το σύστημα εν συγκρίση με τους τεθέντες στόχους. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε κάποια συνοχή. το Stronger and Smarter uh, Information System for Border Security, συγγνώμη για την προφορά μου στα αγγλικά, που καλείται Smart Border, είναι ένα πρόγραμμα πακέτο εφή σύνορα. Πάντα με ανησυχούσε, με ταράζει αυτή η έννοια σύνορα. Ίσως είναι ευκαιρία να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση υπό τον όρο όμως ότι δεν γίνονται παράλληλες κινήσεις ε, επί ολοκληρωμένων συστημάτων, συστημάτων που θεωρούνται ταγμένα. Αν δούμε την πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την ενίσχυση των στοιχείων στα σύνορα, υιοθετήσαμε το PNR. Παράλληλα, χάρη στην άποψη πολλών, έχουμε και το πακέτο για την προστασία των δεδομένων. Αλλά πρέπει να έχουμε και συνοχή. Θέλουμε να τροποποιήσουμε το Eurodac, Μιλάμε για την εξέταση αναγκαιότητας να αναθεωρηθεί το VIS. Δεν τα βλέπω ξεκάθαρα. Όταν λέτε να καλύψουμε τα κενά και τα ρήγματα, θα ήθελα να είναι προς το όφελος ε, υπέρ μάλλον της προστασίας των δεδομένων που αφορούν τους πολίτες καταρχάς. Ευχαριστώ κύριε Βερζιά, πάντα καλό και χρήσιμο να ζητάτε το λόγο, κυρίως αν δεν το ήξερα ότι ήσασταν σκιώδης. Η κυρία Ιντφελτ, δεν είμαι σκιώδης, όμως, ανησυχώ λίγο για όλα αυτά. Όχι διότι είμαι αντίθετη με την αρχή, όχι. Αλλά αν δείτε το όλο ιστορικό του θέματος υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Υπήρχε προκάτοχος της προτάσεως, προηγούμενο. Και η δικαιολογία για την παλιά πρόταση ήταν ότι θέλαμε να εντοπίσουμε εκείνους που έμεναν μετά την εκπνοή της θεωρησής τους και μετά κινηθήκαμε να κάνουμε κάτι άλλο ή θέλουμε να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο των ξένων μαχητών. Μετά υπάρχει και κάποια αλλαγή λειτουργίας ε, σε κάποια από τα στοιχεία που αναφέρατε, το Eurodac, το οποίο όταν το αποφασίσαμε πριν από πολλά χρόνια μας είπαν ότι είναι μόνο για διαπίστωση ταυτότητας, εξεκρίβωση ταυτότητας, τίποτα άλλο. Θυμόσαστε? Καμία φορά αξίζει να θυμάται κανείς. Σιγά σιγά δηλαδή χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Ε, ε, αναφερθήκατε επίσης και στο Ευρωπαϊκό Σύστημα ΕΦΤΑ, ηλεκτρονική έγκριση για ταξίδια. Ε, στον προηγούμενο γύρο, όταν μιλούσαμε για την πρώτη πρόταση για τα αφή σύνορα, είχα θέσει μια ερώτηση και είπα, οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν σύστημα εισόδου-εξόδου και από ό,τι γνωρίζω εξακολουθούν να έχουν πρόβλημα να το εφαρμόσουν πλήρω. Τι μα κάνει να πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Θα ήθελα να μου πείτε κάποια πράγματα περισσότερα και είναι ταμπού αυτό. Τα οικονομικά συμφέροντα. Αυτά τα συστήματα πρέπει να κατασκευαστούν από επιχειρήσεις. Εγώ είμαι φιλελεύθερη. Είμαι υπέρ φιλελεύθερης φιλελεύθερη οικονομία. Να βγάζουν λεφτά οι εταιρείε, εντάξει. Ποια συμφέροντα υπάρχουν, τι παίζει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σε επαφή με εταιρείε του τομέα. Διότι έχουν την τεχνογνωσία, έτσι δεν είναι. Θα ήθελα να μου πείτε Λοιπόν, ποιες εταιρείε ε, ψάξατε, με ποιους ήρθατε σε επαφή, τι συστάσεις δόθηκαν, τι οικονομικά ποσά τίθενται, γιατί ποσά μιλάμε. Ο κ. Κορίος θα το επιβεβαιώνει, αρχικές εκτιμήσεις του κόστους των προγραμμάτων ε, δεν είναι και απόλυτα ακριβή. Το SIS τελικά κόστησε εξαπλάσια από τις προβλέψεις. 8 φορέ παραπάνω από ό,τι προβλεπόταν. Και δεν βλέπω τεράστια συστήματα πληροφορικής που ήταν επιτυχή και παρέμειναν στα όρια τα οικονομικά που είχαν προβλεφθεί. Καταρχήν δεν έχω πρόβλημα. Αλλά λέω με κάποια σιγουριά ότι μπορώ να είμαι διστακτική όσον αφορά αυτά που υπόθηκαν. έχω αμφιβολίες. Ευχαριστώ. Η κυρία Λάουριστεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να συνεχίσω στο ίδιο πνεύμα. Λοιπόν, προστασία δεδομένων και τη νέα κατάσταση που κρατεί για αυτά. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε ποια στοιχεία χρησιμοποιούνται, πώς συλλέγονται και πρέπει να είναι περιορισμένου σκοπού η επεξεργασία των δεδομένων. Άρα πρέπει να συζητήσουμε τι είδους στοιχεία χρειαζόμαστε για να έχουμε αυτό το χώρο, τον κοινό χώρο ασφαλείας. Έχουμε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που εξελίσσονται, δημιουργούνται νέα καθήκοντα, έχουμε υποργανισμούς, Europol, Eurodac, Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή. Όλοι οι φορείς χρειάζονται στοιχεία. Άρα πρέπει να καταλάβουμε για λόγους ασφαλείας ποια στοιχεία χρειαζόμαστε. θα έχουμε μια ενιαία βάση ή εναρμονισμένες βάσεις δεδομένων κρατών μελών. Δεν κάνει μεγάλη διαφορά στο κάτω-κάτω. Θα πρέπει να έχουμε δείκτες που χρειάζονται για τη συλλογή των στοιχείων και από την άλλη πλευρά να τηρούνται αυτά που αποφασίσαμε. Ασφάλεια, προστασία της ιδιωτικής ζωής, προστασία του ατόμου, ε, ό,τι είναι στην οδηγία και στους κανονισμούς, όχι μόνο στην οδηγία. Οδηγία σημαίνει είναι κάτι που αφορά κάτι που συνδέεται άμεσα με κάτι με, που συνδέεται με το έγκλημα. Αυτό αναφέρει η οδηγία. Αλλά η εκτοφυλακή δεν συνδέεται με κάποιο έγκλημα. Εφηή ε, σύνορα δεν συνδέεται με έγκλημα. Ε, πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνουμε. Στο γενικό πλαίσιο. Το να δημιουργούμε αλληλουχία πρωτοβουλειών ε, είναι κάτι που οδηγεί σε σύγχυση. Πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι ο απότερος σκοπός, ποια είναι τα όρια, τι είδου στοιχεία χρειαζόμαστε. Μας λείπουν κάποια στοιχεία. Κοιτάξτε, για τους πρόσφυγες τι έχουμε. Τεράστια κένα, έλλειψη στοιχείων για τους πρόσφυγες. Δεν συλλέγονται. Θα τα χρειαστούμε. Μιλάμε για ένταξη. Αλλά δεν έχουμε στοιχεία. Ε, ποιο θα συλλέγει, για ποιο σκοπό, τα ανθρώπινα δικαιώματα, πώς προστατεύονται. Θα πρέπει να συζητήσουμε αυτό το θέμα ε, των στοιχείων πιο μερός. Κυρία Λόριστεν. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ όλους για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις περισσότερες από αυτές. σχετικά με την προστασία των δεδομένων και τους ε, περιορισμούς ως προς το σκοπό. Η πρόταση σχετικά με το σύστημα εισόδου-εξόδου και το ε, υπάρχον σύστημα είναι συμβατά με τον κανονισμό για την προστασία δεδομένων και το πολύ αυστηρό πλαίσιο που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι λεπτομέρειες, πιστεύω, είναι για ε, να ολοκληρωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο και θα σας παρουσιαστούν φυσικά στην Επιτροπή. Ε, σας εγγυώμαι όμως ότι θα ε, εφαρμοστούν όλες οι ασφαλιστικές δικλίδες και θα ισχύουν οι αρχές της ιδιωτική, ιδιωτικότητας κατά, την, κατά το σχεδιασμό του συστήματος. Τώρα, για τις νέες προτάσεις που σχεδιάζουμε και για το ότι παράλληλα σκοπεύουμε να συστήσουμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων. Καταρχάς, η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα ασχοληθεί με συγκεκριμένες πτυχές διαλειτουργικότητας. Θα αναλύσει το ενδεχόμενο ή την ανάγκη να ε, επεκτείνουμε τη θελητουργικότητα. Αυτό συμπεριλαμβάνεται στην ανακοίνωση. Επίσης, δεν καλύπτονται κάποιοι τομείς. Ε, σωστά υπάρχουν κάποια κενά πληροφοριών, για παράδειγμα ταξιδιώτες χωρίς θεώρηση που φτάνουν σε εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουμε πληροφορίες μέχρι την άφηξή τους. Αυτό θεωρούμε κενό στην πληροφορία για τη... τους ελέγχους στα σύνορα. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πρόθεση να αναλύσει την αναλογικότητα ε, και να προτείνει τη δημιουργία ενός συστήματος έγκρισης ε, ταξιδιού. Και για τον ίδιο σκοπό έχουμε την υποχρέωση να αναλύσουμε και να αναθεωρήσουμε τους διάφορους κανονισμούς σχετικά με το SIS, το EU το VIS. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τέλος περίπου της διαδικασίας αξιολόγησης για τους περισσότερους κανονισμούς. Επίσης, έχουμε τοπίσει την ανάγκη να προτείνουμε τροποποιήσεις για κάποιους από αυτούς τους κανονισμούς έτσι ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία των υπηρεσιών. Τώρα, σχετικά με την εντολή και την χρηματοδότηση και τους περιορισμούς του EU Λίζα, υπάρχουν συστήματα γι' αυτό. Ποιότητα δεδομένων. Όπως ανέφερα στην αρχή, χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι τα συστήματα που έχουμε χρησιμοποιούνται με τρόπο αποτελεσματικό και οι πληροφορίες που καταγράφονται σε αυτά τα συστήματα είναι συμβατές με τον κανονισμό. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, γι' αυτό πρέπει να είναι συμβατή με ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές. Οι πληροφορίες που υπάρχουν στο σύστημα μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση συγκεκριμένων ατόμων, γι' αυτό πρέπει να ε, διαχειριστούμε τα δεδομένα αυτά με τον σωστό τρόπο. Είναι επομένως για εμάς αναγκαίο να παρακολουθούμε την ποιότητα των δεδομένων στο EU Lisa, έτσι ώστε να ε, δούμε εάν είναι εφικτό αυτό, αυτή η χρήση που προβλέπουμε. Τώρα, σχετικά με την κεντρική βάση δεδομένων. Ναι, χρειάζεται ένα κεντρικό αποθετήριο, μια κεντρική τράπεζα δεδομένων. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αξιολογήσει η ομάδα υψηλού επίπεδου εμπειρογνωμόνων και είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος που έχουμε. Είναι ο τέταρτος στόχος. Ο πρώτος στόχος είναι δηλαδή να χρησιμοποιηθεί ένα νέο σύστημα έρευνας. Δεύτερος, η διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων. Τρίτον, ε, ο, η καλύτερη χρήση και βελτίωση του ΕΦΙΣ, του συστήματος για τα δεκτυλικά αποτυπώματα και εάν χρειαστεί να υπάρχει η δυνατότητα για μια πιο ενοποιημένη βάση δεδομένων. Όταν δηλαδή καταχωρείς, δεδομέ, δεδομένα σε μία βάση δεδομένων ε, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι υπάρχουν και παραβιάσεις. Κάθε πληροφορία που ε, καταγράφεται, καταγράφεται για ένα συγκεκριμένο σκοπό και αυτό θα φαίνεται. Και οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και σύμφωνα πάντα με την προστασία δεδομένων. Και θα ακολουθεί το σκοπό για τον οποίο ε, επεξεργάζεται τα δεδομένα. Ε, δεν δια Κινδυνεύουμε λοιπόν την ασφάλεια των δεδομένων με το να καταγράφονται όλα σε μία βάση δεδομένων. Τώρα, οι διάφοροι κανόνες σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων θα ε, διέπουν την εκάστοτε χρήση τους. Η ενοποίηση δηλαδή των συστημάτων δεν σημαίνει ότι θέλουμε να αλλάξουμε ε, τους κανόνες που θα διέπουν τη διατήρηση, την επεξεργασία και τον τρόπο που θα χρησιμοποιούνται τα δεδομένα. Νομίζω πως ήδη απάντησα για την προστασία των δεδομένων. Η διαλειτουργικότητα, όπως είπα, δεν σημαίνει πως θα ανακατέψουμε τα δεδομένα από τα διαφορετικά συστήματα. Σημαίνει ότι θα εγκρίνεται η χρήση των δεδομένων από ένα άλλο σύστημα. Από το να υπάρχουν δηλαδή διάφορες και πολλές ανταλλαγές δεδομένων ανάμεσα στα διάφορα συστήματα θα υπάρχει δυνατότητα απλοποίησης μιας αναζήτησης έτσι ώστε ένας χρήστης να μπορεί να ε, κάνει παράλληλα ε, πολλές αναζητήσεις και αυτό θα οδηγήσει στη μείωση της ε, κίνησης των πληροφοριών στα δίκτυα και στα εθνικά συστήματα και εδώ εξετάζουμε το ενδεχόμενο να δημιουργήσουμε διαλειτουργικότητα σε ένα κεντρικό επίπεδο ανάμεσα σε όλα τα, αυτά τα συστήματα. Όμως φυσικά θα γίνεται, σεβαστή, ε, θα γίνεται σεβαστό το δικαίωμα πρόσβασης του χρήστη στο σύστημα. Δεν θα αλλάξουν δηλαδή τα δικαιώματα χρήσης. Επίσης, αυτή η διαλειτουργικότητα σε κεντρικό επίπεδο πρέπει να είναι συμβατή με την προστασία δεδομένων και με την ε, σχετική νομοθεσία για μείωση της κίνησης μεγάλου όγκου δεδομένων. Δεν θα αντιγράφονται τα δεδομένα σε πολλά συστήματα ταυτόχρονα. Θα υπάρχει δυνατότητα με μία αναζήτηση να αντλείς από διάφορα συστήματα την πληροφορία που θες. Αυτό θα προβλέπει ο κανονισμός. Θα αποφευθεί δηλαδή το να δημιουργούνται διάφορα, διαφορετικά αντίγραφα δεδομένων σε όλα τα συστήματα. Τώρα, τα δεδομένα που θα συλλέγονται. Η ομάδα πυρογνωμόνων υψηλού επίπεδου, μεταξύ άλλων, θα εντοπίσει όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για να αποφύγουμε το να μην ταυτοποιούνται ορισμένοι ταξιδιώτες. Και με αυτό νομίζω πως απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ και όλους τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους. Θα συνεχίσουμε τώρα την συνεδρίασή μας στις 3 το μεσημέρι και σας εύχομαι καλή όρεξη.